Good afternoon. If everybody can take his or her place. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας σήμερα. Σας καλωσορίζω σε αυτήν τη συνεδρίαση που έχουμε αυτό το απόγευμα της Υποεπιτροπής μας Άμυνας και Ασφάλειας. Η σημερινή μας δημόσια ακρόαση θα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στους προϋπολογισμούς άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνατότητες και ευκαιρίες για κοινέ συμμετοχές και κοινέ προμήθειες. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλοξενουμένους, προσκεκλημένους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αυτό το θέμα. Μία μελέτη έγινε και η επόμενη πρωτοβουλία, μελέτη πρωτοβουλία θα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Με την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, χρηματοοικονομική κρίση που έχει σημαντικέ επιπτώσεις στους προπολογισμού άμυνας, πρέπει να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε το δυναμικό μας, τα στελέχη και τον εξοπλισμό αν θέλουμε συλλογικά ή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο ΝΑΤΟ να εγγυηθούμε τα θέματα ασφάλειάς μας και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις αξίες και τις αρχές μας από απειλές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συνθήκη της Λισαβόνα δίνει αρκετά εργαλεία για την αναβάθμιση της συνεργασίας μας στην άμυνα η πιο απαιτητική αυτή συνιστόσα είναι η συνεργασία. Αλλά πρέπει επίσης να σημειώσουμε τον ε, διευρυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας που θα προαγάγει την Ευρωπαϊκή Άμυνα στην τεχνολογική και βιομηχανική της βάση. Η συνθήκη επίσης αναφέρει ευρωπαϊκό δυναμικό και πολιτική για τους εξοπλισμούς. Αυτές οι νέες πολιτικές σε συνδυασμό με τις αγορές άμυνας και τις μεταφορές τεχνογνωσίας θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την αυτονομία στρατηγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την δική της ικανότητα να υπομίζεται ευθύνες παγκόσμια. Προσωρινά θα πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση των σημερινών δυνατοτήτων που έχουμε οι κοινέ ευκαιρίες που προσφέρονται και οι προμήθειες από το 2007 από αυτή την προσέγγιση τίθενται πολλά ερωτήματα για την διαθεσιμότητα και την κυριαρχία και ελπίζω ότι όλα αυτά τα θέματα θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ένας τρόπος χρήσης των σπανιζόντων πόρων μας είναι να ξεκινήσουμε κοινά προγράμματα με στόχο να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας και εν τέλει θέλει, πρέπει να διασφαλίσουμε αν νέα κονδύλια και νέες δυνατότητες πόρων μπορούν να δημιουργηθούν ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει κάποιες από τις δυνατότητες που χρειάζονται για τις αποστολές υπό την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησαν οι πρωτοβουλίες και δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις ανάγκες της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Με αυτή την ακρόαση θέλουμε να διεξαγάγουμε έχουμε μια κοινή ακρόαση για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ελπίζουμε ότι στο τέλος των συζητήσεων θα έχουμε βρει κάποιες από τις απαντήσεις που αναζητούμε. Η συζήτηση διαρθρώνεται σε δύο βήματα, σε δύο πάνελ. Για το πρώτο έχω την χαρά να να καλωσορίσω τον κύριο Κρίστιαν Μέλινγκ από το Ίδρυμα Επιστήμης ε, ε, και ε, σας στο Βερολίνο και πολιτικής του Βερολίνου που έχει αναλάβει αυτή την ε, μελέτη. Επίσης ε, τον ε, κύριο Μελάης που έχει αναλάβει από πλευράς των Παρισίων μελέτη. Θα επικεντρωθούμε στο πάνελ αυτό στις συνέπειες των δημοσιονομικών περικοπών στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά την απώλεια δυναμικού, στρατιωτικού δυναμικού και την ανάγκη να εξευρεθούν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης. Ξεκινάμε με τον Γερμανό φιλοξενούμενο Δ. Μέλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τεχνικούς λόγους θα παρουσιάσω την παρουσίαση αυτή και θα είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις στη συνέχεια. Uh, Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, αναλάβαμε στο Γερμανικό Ινστιτούτο να κάνουμε μία μελέτη για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης ε, στα θέματα άμυνας της Ευρώπης. Αυτό κάναμε τους τελευταίους μήνες και θα παρουσιάσουμε τα ευρήματα αλλά και κάποια ε, συμπεράσματα. Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε δύο βασικά προβλήματα τα οποία συνέπεσαν τα τελευταία χρόνια. Το ένα αφορά την δημιουργία ικανοτήτων και το δεύτερο είναι η οικονομική κρίση. Η δημιουργία ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αντιμετωπίζει μάλλον τρία προβλήματα τα οποία δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Καταρχάς έχουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια ευαισθητοποίηση αλλά δεν υπάρχουν πόροι από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν φτάσουμε στις ικανότητες υπάρχουν οι εξοπλισμοί. Αυτό είναι ένα θέμα ε, εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ σχετίζονται τα προβλήματα με την ε, βιομηχανική τεχνολογία και τον χώρο εργασίας. Το τρίτο πρόβλημα δημιουργείται από την έλλειψη αν θέλετε σύνδεσης και επαφής ανάμεσα στα, στους, στα διάφορα, διάφορους οργανισμούς, διάφορους πόρους γιατί δεν συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό δεδομένο. Τώρα όμως έχουμε και ένα επιπλέον πρόβλημα που είναι η οικονομική κρίση. Και όπως συνειδητοποίησαμε από τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε δύο δεκαετίες οικονομικής κρίσης. Καταρχάς είχαμε μαζική μείωση των πόρων και αυτή θα διευρυνθεί τους τις επόμενες δεκαετίες. Δεύτερον ε, υπάρχουν ε, περιορισμένοι πόροι και περικοπές που διαφέρουν βέβαια από χώρα σε χώρα. Παρόλα αυτά υπάρχουν δημοσιονομικές περικοπές, 30% για τις μικρές χώρες, ε, για τις μεσαίες χώρες 10 και 15% και οι μεγάλες χώρες ε, γύρω στο 8%. Προσπαθούν δηλαδή κάποιες χώρες να ξεφύγουν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά όπως ε, ε, έχει παρουσιάσει η Κομισιό, τα επόμενα 20 χρόνια θα ε, ξοδέψουμε στην Ευρώπη 1% του ΑΕΠ μας για να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω χρέη. Πιστεύουμε ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορέσει να ε, διευρύνει ή να διατηρήσει τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Το επίπεδα ε, φιλοδοξίας ε, αν θέλετε της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης παραμένουν ως έχουν παρόλα αυτά, επισήμως τουλάχιστον παρόλα αυτά de facto γίνεται μια εξειδίκευση το Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια και η Γερμανία έχουν, και οι κατοχώρες έχουν περιορίσει το επίπεδο φιλοδοξιών και υπάρχουν περικοπές ε, και όσον αφορά ε, τον, και τους εξοπλισμούς και, τις, και το προσωπικό. Υπάρχει επομένως και μία εξειδίκευση de facto, αλλά υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες δημοσιονομικές περικοπές. Το πρόβλημα είναι ότι ε, ούτε εμεί ούτε τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να ε, ξεκαθαρίσουν γιατί δημιουργούνται αυτά τα κενά ικανοτήτων. Όσον αφορά το κόστος του προσωπικού, το 5% ίσως και παραπάνω των αμυντικών δαπανών αφορούν το προσωπικό αλλά εδώ δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν δυνατότητες για εξοικονόμηση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Όσον αφορά τους εξοπλισμούς έχουμε ένα αυξανόμενο κενό ανάμεσα σε αυτούς που εξυγχρονίζουν με αργό ρυθμό και αυτούς που κάνουν περικοπές στις προμήθειές τους. Τώρα, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, εξετάζονται νέες αγορές έτσι ώστε να ε, προλάβουμε κάποιες ε, περικοπές ή ίσως καθυστερούμε κάποια νέα project. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν σαν στόχο να διατηρήσουν τις εθνικές αμυντικές τους βιομηχανίες. Η μελέτη την οποία κάναμε, καμιά φορά την ξεπερνάνε τα γεγονότα. Γιατί έχουμε πληροφορίες ότι ολοένα και περισσότερα στρατεύματα αποσύρονται από τις ε, διεθνείς αποστολές, άρα βλέπουμε ότι δεν γίνεται μόνο μία αναδιάρθρωση των εθνικών προτεραιοτήτων, αλλά υπάρχει και μία απομάκρυνση αν θέλετε από τις ε, διεθνείς ε, δεσμεύσεις μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ε, το pooling και sharing, δηλαδή μια κοινή εκμετάλλευση, είναι το μότο το οποίο επικρατεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές διμερείς ή πολυεθνικές πρωτοβουλίες Υπάρχουν τα πρώτα δείγματα για μια νέα πολιτική διαδικασία που ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω ή μπορεί να πρόκειται και για ένα πρόβλημα που θα αρχίσει να αντιμετωπίσει η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θα δούμε ποιο, είναι το, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Έχουμε την πρωτοβουλία της Γάνδης, ε, η οποία έχει σαν στόχο να ξεπεράσει τις γραφειοκρατίες. Αυτή τη στιγμή η, η αντιμετώπιση είναι κάπως μεικτή. Έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι, ε, θέλουν να κάνουν κάτι, έχουμε τους απεσιόδοξους και έχουμε και τους ειδικού. Θα πρέπει να δούμε τις πρόσφατες εξελίξεις όπου βλέπουμε να υπάρχουν 100 περίπου projects για κοινή εκμετάλλευση και χρήση, και χρήση των ικανοτήτων. Ο κανόνας είναι το bottom-up, από κάτω προς τα πάνω δηλαδή. Ε, έχουμε διμερείς συμφωνίες ε, γύρω στο 20%, διμερεί project γύρω στο 20% Ούτως ή άλλως βέβαια τα, τα μεγαλύτερα project αφορούν το ΝΑΤΟ και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ο Τόμας Μάουλινγκ έχει κάνει μια εξαιρετική ε, μελέτη για τα θέματα αυτά, άρα θα τα συζητήσουμε αργότερα. Και επανέρχομαι εδώ στην, ε, στην αρχή ε, της παρουσίασής μου που αφορά την τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς δηλαδή την δημιουργία ικανοτήτων και την οικονομική κρίση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς την ύπαρξη και τη φύση του προβλήματος, άρα δεν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση. Ε, γίνονται σπασμωδικές κινήσεις. Βέβαια, με την οικονομική κρίση εμφανίστηκαν τα διάφορα προβλήματα που είχε η αμυντική πολιτική, ε, οδήγησε σε μια επιτάχυνση των περικοπών, Δεν ξέρουμε βέβαια αν είμαστε μάρτυρες ε, ε, ενός αργού θανάτου της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα και να δημιουργήσουμε ε, μια νέα πολιτική ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη. Είδαμε τι έγινε και στην Λιβύη τον τελευταίο, ε, ε, τον τελευταίο καιρό οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα είναι στο μέλλον διαθέσιμες για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ή τα κράτη-μέλη είναι ικανά να προσφέρουν ασφάλεια. Επίσης, η οικονομική κρίση αυτό το οποίο έκανε είναι να ενδυναμώσει μια γενικότερη τάση ότι δεν έχουμε πλέον χρόνο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδυαστεί η βιομηχανική διάσταση και η διάσταση ικανοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ούτως ή άλλως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δούμε μακροπρόθεσμα. Μεσοβραχυπρόθεσμη λύση δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τα ε, εξής βήματα. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τις ικανότητες να ικανοποιήσουμε, να υπηρετήσουμε τις φιλοδοξίες ε, τις οποίες έχουμε θέσει. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πρώτο βήμα. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις εξελίξεις, ε, θα πρέπει να επενθυμίσουμε τα κράτη-μέλη ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, ε, τι έχουν προσυπογράψει στις συνθήκες. Τώρα, σε επίπεδο θεσμών θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Θα πρέπει να και οι υπουργοί σε πολιτικό επίπεδο να ευαισθητοποιηθούν. Επίσης θα πρέπει να παίξουν έναν ρόλο και Υπουργοί Οικονομικών. Γιατί ο ρόλος τους σε περίοδο, στην περίοδο λιτότητας στην οποία ζούμε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τα project κοινής ε, των κοινών επενδύσεων. Θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με τον ΝΑΤΟ. Τώρα, όσον αφορά τις ικανότητες, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τα, τις μαχητικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι σαν μονάδα πολεμική αν θέλετε, αλλά σαν ένα εργαστήριο. Δηλαδή θα πρέπει να διευρύνουμε το μέγεθος αλλά και την, και τον, την χρήση, τον χρόνο χρήσης αυτών των ομάδων μάχης Επίσης, θα πρέπει να εξάγουμε τα διδάγματά μας από όλες τις αποστολές τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο καιρό και όσον αφορά τους εξοπλισμούς για την ε, Ευρωπαϊκή Άμυνα θα θέλαμε να προτείνουμε κάποιο, ένα γενικότερο στόχο για το 2030 Καταρχάς δηλαδή θα πρέπει να εντοπίσουμε την, ε, τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες ε, της πολιτικής μας. Θα πρέπει επίσης να συντονίσουμε τις βιομηχανικές μας πολιτικές και προτεραιότητες και να εναρμονίσουμε τον κύκλο προμηθειών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε τώρα στον δόκτορα Μπελέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά για να μην ε, κατακρεουργήσω την αγγλική γλώσσα. Βέβαια μετά από όσα είπε ο κύριος Μέλινγκ ε, είναι δύσκολο να πάρω εγώ το λόγο, αλλά θέλω να πω ότι ε, και εγώ έχω αναλάβει τη διεξαγωγή μιας μελέτης στο πλαίσιο της Ένωσης Eurodefense που θα τη δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις αμυντικές προσπάθειες μεταξύ Ευρώπης και ΕΠΑ Στόχος είναι να δούμε πώς εξελίσσονται οι δαπάνες στον τομέα της άμυνας. Είναι πιο πολύ πανεπιστημιακή η προσέγγιση και όχι τόσο ε, επαγγελματική. Βλέποντας ε, τις δημοσιονομικές εξελίξεις που είτε έχουν ανακοινωθεί είτε έχουν αποφασιστεί, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί οι βασικότερε τρει χώρε που αντιπροσωπεύουν το 60% των αμυντικών ε, δαπανών έχουν ε, ακολουθήσει τώρα τη λογική περιστολή των αμυντικών δαπανών και οι εκτιμήσει είναι πολύ σημαντικέ λόγω τη οικονομική κρίση και των επιπτώσεων που είχε στα δημόσια οικονομικά. Βλέπουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 8% μέσα σε 4 χρόνια θα μειωθούν οι αμυντικέ δαπάνε ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μείνουν γύρω στο 2% του ΕΠ. Στη Γαλλία Σήμερα γίνεται λόγος για μείωση κατά 3,5 δις μέχρι το 2013 με ε, αναθεώρηση ε, επιταχύρω των αποτελεσμάτων που είχαν παρουσιαστεί. 8,3 δις θα είναι ο προπολογισμός στη Γερμανία μέχρι το 2014. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ η άμυνα είναι μια σημαντική θέση του προπολογισμού στα κράτη-μέλη, ήδη βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν προσπάθειες συνένωσης πόρων σε σχέση με τις ΗΠΑ που έχουμε 4% ποσοστό του ΑΕΠΑ, ίσως και περισσότερο ε, αν λαμβάνουν υπόψη επιχειρήσεις Αφγανιστάν και Ιράκ Ε, σε εμά μιλάμε για 1,7% κατά μέσο όρο. Άρα, ποια είναι η δική μας θέση απέναντι στι. ΕΕ. Υπάρχουν κάποια κατόφλια ενδεχομένω ε, στι αμυντικές ε, δαπάνε. Ίσως ε, θα μπορούσε κανείς να δει ότι δεν υπάρχει μια γραμμική προσέγγιση και βλέπουμε ότι μειώνονται οι αμυντικές δυνατότητες και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης. Και βλέπουμε και τι γίνεται και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Παρά τις υψηλές αμυντικές δαπάνες δεν είναι υψηλές οι αμυντικές δυνατότητες των κρατών μελών. Μακροπρόθεσμα τώρα, και αν δούμε το 96 είχε γίνει και από εκεί και πέρα, οι αμυντικοί προπολογισμοί και ιδίω οι επενδυτικοί προπολογισμοί είχαν τελματώσει για μια 15 περίπου. Άρα, ναι μεν αυξάνονται οι προπολογισμοί, σε όταν αφορά την αγοραστική τους δύναμη έχουν τελματώσει, ε, έχουν παραμείνει στάσιμοι. Και αυτό είναι πρόβλημα, όπως βλέπουμε, διότι το κόστος των εξοπλισμών αυξάνεται, και η τάση μακροπρόθεσμη που δείχνουν και οι οικονομικές μελέτες είναι ότι το κόστος των εξοπλισμών αυξάνεται κατά 5 ε, με 7% το χρόνο και αυτό σημαίνει ότι αν οι προπολογισμοί ακολουθήσουν τον πληθωρισμό τότε η αγοραστική δύναμη μειώνεται προοδευτικά. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ε, τις εξοπλιστικές βλέπουμε ότι είναι σταθερή η τάση γύρω στα 20 δις για το Ηνωμένο Βασίλειο, 8 ε, δις για τη Γερμανία, 5 δις για την Ιταλία, 3 δις για την Ισπανία. Μόνο η Γαλλία ε, στα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι μέχρι το 2003 είμαστε στα 12 δις και έχουμε αυξήσει, έχουμε φτάσει στα 16 δις τα τελευταία χρόνια. Επειδή όμως ανακοινώθηκαν περιστολές, βλέπουμε ότι θα μειωθούν και στη Γαλλία οι αμυντικές δαπάνες. Δεύτερον, Πέραν αυτή τη ε, στάσιμης προσπάθεια βλέπουμε ισχυρότερε πιέσει μείωση των δημοσίων δαπανών. Όπως βλέπετε στις χώρες του ΟΣΑ το δημόσιο έλλειμμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. 98 έως 2007 ήταν γύρω στο 2% του ΑΕΠ. Έχει γίνει 8% το 2009 περίπου. Βλέπουμε ότι οι χώρες της Ευρωζώνης δεν έχουν βέβαια τόσο πολύ μεγάλο έλλειμμα, αλλά παρόλα αυτά έφτασε κάποια στιγμή και το 6,3% συγκεκριμένα το 2010. Οι ευρωπαϊκέ χώρε, βέβαια, σε σχέση με άλλε χώρε, έχουν πολύ μικρότερα περιθώρια ελιγμών λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που προποθέτουν μια ε, ισορροπία, μια ισοσκέληση στου προπολογισμού. Άρα εδώ βλέπουμε ότι για να ε, αποκαταστήσουμε την ισορροπία και να φτάσουμε στους αρχικούς δείκτες ε, πρέπει να ασκηθεί πίεση στις χώρες για να έχουν ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή λιγότερες πάνε σε σχέση με τα έσοδα. Όλα αυτά θα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, ιδίω βλέποντα κανεί τι στατιστικέ ε, περί, δημοσίου χρέους. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πολύ το χρέος, ε, έχει σχεδόν ε, εκτοξευθεί. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί για να επανέλθουμε στους αρχικούς δείκτες. Όπω είπε και ο Δόκτωρ Μέλλιν, τώρα, η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι έχουμε φτάσει στα όρια ε, τη μείωση των αμυντικών ε, επενδυτικών προσπαθειών. Βλέπουμε τι γίνεται στη Λιβύη, παραδείγματο χάρη. Βλέπουμε ότι χωρί αμερικανική στήριξη οι ευρωπαϊκέ χώρε δεν θα μπορούσαν να παρέμβουν. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα και μόνο αν δει κανεί τη χρήση των πυράβλων από τι Αμερικανικέ δυνάμει, βλέπουμε ότι το σύνολο των πυράβλων που εκτοξεύονται από τι Αμερικανικέ δυνάμει αντιστοιχούν, μέσα σε μια εβδομάδα, αντιστοιχούν στο σύνολο ενό μείζων ε, προγράμματο ε, πυραυλικού. Το Σκάλπελ Ναβάλ, παραδείγματο χάρη στη Γαλλία, όπου είμαστε στου 200 συνολικά πυράβλου. Σήμερα Βέβαια, καταφέραμε να διατηρήσουμε το σύνολο των προγραμμάτων και των δυνατοτήτων, αλλά είναι τόσο χαμηλό αυτό το επίπεδο που ουσιαστικά δεν έχουμε πραγματικές αμυντικές ε, δυνατότητες ε, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε τη δυνατότητα, ότι έχουμε δύναμη παρέμβαση και μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά αν τελικά ε, μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα, τι, περί τίνος δυνατότητας μιλάμε επί τη ουσία Και αν δει κανεί και το διασκορπισμό και τον κατακαιρματισμό και των δαπάνων και των προγραμμάτων, ε, μπορεί να συναγάγει τα δεόντα συμπεράσματα. Ίσως λοιπόν κάθε μη προγραμματισμένη δαπάνη στο μέλλον καταστεί αδύνατη, ανέφικτη και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και από πλευράς άμυνας και από πλευράς ε, δυνατότητας παρέμβασης ή επέμβασης. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την ψαλίδα 5 με 7% αυξάνουν οι πρώτες ύλες σε μακροπρόθεσμα για τα βασικότερα ε, προγράμματα και έχουμε ένα είδος ε, ψαλίδας. Έχουμε κάποιους πόρους που διατηρούνται σε ένα σταθερό όμως επίπεδο, σχεδόν σταθερό και απ' την άλλη έχουν αύξηση του υλικού ε, και των εξοπλισμών. Και έτσι καθίσταται όλο και πιο δύσκολη αγορά εξοπλισμών. Αν οι δημοσιονομικές τάσεις συνεχιστούν κατά αυτόν τον τρόπο, όπως ήταν στη δεκαετία του 1990, το Πεντάγωνο ε, δεν θα μπορεί το 2030 να αγοράσει παρά ένα μόνο μαχητικό αεροσκάφος. Ε, μήπως τελικά ε, αυτό συμβεί στην Ευρώπη. Θα ήταν κρίμα. Επόμενα θέματα. Πρώτο ερώτημα. Είναι εύλογο να έχουμε ε, μία προσέγγιση περιστολής δημοσίων δαπανών. πρέπει να προηγηθούν οι αμυντικές δαπάνες σε βάρος άλλων Νομίζουμε ότι όλα τα Υπουργεία σε όλες τις χώρες πλήττονται από περικοπές, αλλά δεν έχουν όλα τα Υπουργεία τους ίδιους στόχους, αλλά ούτε και τα ίδια μέσα. Αν δούμε την άμυνα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι αυτό είναι το βασικό Υπουργείο που δαπανά σε κεφάλαιο, το Υπουργείο Άμυνας. Άρα είναι σημαντικός ο στόχος. Δεύτερο, δεύτερο ερώτημα, πρέπει τη μείωση των ε, αμυντικών δαπανών ε, να την διαχειριστούμε εντός των προπολογισμών και θα πρέπει να δει κανείς την ιστορία, δηλαδή τέλος ψυχρού πολέμου. Τι γινόταν τότε. Στην Ευρώπη διατηρήθηκαν οι κοινωνικές, θα έλεγα, στρατιωτικές δαπάνες, όχι δαπάνες προσωπικού, σε βάρος επενδυτικών δαπανών θυσιάστηκαν δηλαδή πρώτα απ' όλα ε, τα πυρομαχικά, η έρευνα και η ανάπτυξη και μετά οι επενδύσεις. Εάν δούμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ, όλοι οι προπολογισμοί μειώθηκαν, αλλά η μείωση ε, στην ε, περίπτωση της ε, άμυνας ε, και της ε, έρευνας και ανάπτυξης ήταν δύο φορές μικρότερη. Άρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό. Τρίτο ερώτημα πρέπει να λέμε υπόψη κάποιο επίπεδο ε, κάτω φλοιού λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και του μεγέθους της παραγωγής. Αν δούμε εδώ τις βιομηχανικές χώρες για μια δεδομένη τεχνολογία έχουμε ένα δεδομένο μέγεθος αγοράς για να υπάρχει και η βιώσιμη παραγωγή. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη το κατόφλι βιωσιμότητας ε, πώς ορίζεται σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να τεθεί αυτό το ερώτημα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα με συνεργασίες, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το κατόφλι κάποιες φορές, ε, αυτό το ταβάνι, αν θέλετε, η οροφή ε, γίνεται πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την υπερβούμε. Όπω έλεγε ο κύριο Μέλινγκ, λοιπόν, ουσιαστικά η κρίση δεν δημιούργησε τα προβλήματα, αλλά τα αποκάλυψε βλέπουμε ότι οι αμυντικές προσπάθειες έχουν διαβρωθεί και αυτό είχε συγκαλυφθεί λόγω των οικονομικών και νομισματικών προβλημάτων. Άρα τώρα πλέον έχοντας τα προβλήματα μπροστά μας πρέπει να προχωρήσουμε σε λύσεις. Σε δύο άξονες ίσως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε οικονομικά, ένας εγκάρσιος και ένας οριζόντιος άξονας θα έλεγα. πρώτος άξονας που λαμβάνει ακριβώς αυτά τα κατόφλα υπόψη είναι να βρούμε τη σωστή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα προσπάθειας η αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής άμυνας δεν είναι γραμμική σε σχέση με το επίπεδο των δαπανών. Αν μειώσουμε λίγο τις αμυντικές δαπάνες θα έχουμε κλιμάκους, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα κλίμακας. Δηλαδή θα δαπανούμε μεν χρήματα, αλλά η αποτελεσματικότητα θα μειώνεται πολύ σημαντικότητα σε σχέση με τη μείωση του ίδιου του επίπεδου των δαπανών. Και αυτό το βλέπουμε θα είναι εκθετική δηλαδή. Το βλέπουμε και στο πλαίσιο των ε, επενδυτικών δυνατοτήτων, στα νέα προγράμματα ή στις ε, δυνάμεις ε, που μπορούν να αναπτυχθούν. Αν λοιπόν η αγορά δεν ε, μπορεί πλέον να διατηρήσει εν φορέα ή αν δεν μπορεί κάποιο κράτος να εξοπλίζεται μόνο του, θα πρέπει το μέγεθος της αγοράς να αλλάξει. Ο κ. Μέλινγκ είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινή εκμετάλλευση, συνένωση προσπαθειών, ώστε τελικά να βρούμε τη σωστή κλίμακα που θα είναι προσαρμοσμένη στην παραγωγή. Και αυτό ίσως να μην είναι απαραίτητα μια κλίμακα 27 ε, κρατών μελών. Ίσως θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιες χώρες μόνο. Και έτσι ενδεχομένω θα μπορούσε να διατηρηθεί και ο ανταγωνισμό. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα λογική, γιατί ίσω στον μονοπόλιο να μην είναι και καλύτερη απάντηση όταν έχουμε προβλήματα αποτελεσματικότητα. Το σημαντικό εδώ είναι πάντω στην Ευρώπη να διατηρηθεί η δυνατότητα παραγωγή. ώστε η Ευρώπη να είναι σε θέση να αποφασίζει και να βρά από μόνη της. Δεύτερη διάσταση. Και βραχυπρόθεσμη και έτσι με ένα πιο βαθύ προβληματισμό αν θέλετε Οριζόντιος άξονας είναι να δούμε τις σχέσεις μεταξύ κράτους βιομηχανίας. Σήμερα έχουμε ένα βιομηχανικό μοντέλο που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη λογική της δρομολόγησης των προγραμμάτων. Ξεκινάμε λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα για να διατηρηθούν κάποια μελετητικά γραφεία και για να δημιουργηθεί μελλοντική αγορά. Για 50 χρόνια λειτουργήσε αυτή η λογική. Όταν ολοκληρωνόταν η ανάπτυξη ενό ε, προγράμματο και περνάγαμε στην παραγωγή, περνούσαμε στην επόμενη γενιά προγραμμάτων. Σήμερα όμω φτάνουμε στα όρια του μοντέλου αυτού γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε για νέα προγράμματα. Άρα, η λήψη, μάλλον για να μην έχουμε αυτή τη λογική, μήπως θα έπρεπε να αναδιοργανώσουμε τις σχεσεις κράτου κράτους-βιομηχανίας. να διατηρήσουμε τις ε, δυνατότητες και να έχουμε και μια κοινή προσπάθεια μεταξύ χωρών, κοινή εκμετάλλευση δυνατοτήτων. Θα μπορούσαμε ε, με την υποστήριξη παραδείγματος, αν έχουμε κοινή στήριξη, στην προσφορά δηλαδή να έχουμε ε, το pooling and sharing αφού έχουμε πρόβλημα με τη ζήτηση. Βρετανική στρατηγική του 2005 ε, νομίζω ότι ανοίγει ενδιαφέροντες ορίζοντες και ίσως θα έπρεπε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και να δούμε πώς μπορούμε να συνενώσουμε κάποιους πόρους, κάποια μέσα, χωρίς όμως κατά να υπάρχουν και κοινά προγράμματα. Βλέπουμε λοιπόν ε, τις δημοσιονομικές εξελίξεις που δείχνουν ότι χρειάζεται να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της οικονομικής κρίσης. και πρέπει να γίνει επένδυση και στον τομέα τη ε, ζήτηση και στον τομέα τη προσφορά, αλλά πρέπει οι συμβαλόμενοι διάφορε πλευρέ να συμφωνήσουν μεταξύ του. Και ολοκληρώνοντα, θα πω ότι η αμυντική βιομηχανία βασίζεται σε μια εταιρική σχέση μεταξύ κράτου και βιομηχανία, θα ήταν ίσω πιο ε, χρήσιμο να δούμε μια προσαρμογή αυτή τη εταιρική σχέση σε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σα ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε συζήτηση για περίπου ένα μισάωρο μετά από το πρώτο πανέλ. Ξεκινάμε με εσάς κυρία Δούμες, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο και μου, μας αναφέρατε αυτά τα πράγματα. Όχι ότι δεν τα γνωρίζαμε, αλλά είναι σημαντικά να λέγονται αυτά ξεκάθαρα και σταράτα. Γιατί πραγματικά έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι δεν ανταποκρινόμαστε στους στόχους μας, δεν πετυχαίναμε τους στόχους μας και ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση ακόμα λιγότερο. Και αν θέλουμε να έχουμε ένα υπόδειγμα των ελλείψεων και ελληματικής μας κατάστασης, αυτό το υπόδειγμα είναι η Λιβύη. Διότι όλες οι απαιτήσει για την Ευρώπη που θα έπρεπε να λειτουργήσει η Ευρώπη υλοποιώντα το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε η Ευρώπη να δώσει τα ενία στο ΝΑΤΟ και μια και οι Αμερικανοί πίστευαν ότι ήταν ευρωπαϊκή δουλειά κυρίως που έπρεπε να γίνει και αυτό παρότι αυτό το κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο από την αρχή κιόλα ζήτησε να υπάρξει μια αποστολή της CSDP για την υλοποίηση του εμπάργου όπλων που είχε αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το πρόβλημα είναι ότι με την έλλειψη πόρων και δυνατοτήτων λόγω της οικονομικής κρίσης Υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις όμως παρόλα αυτά σε σχέση με τις ανάγκες για την ασφάλεια που είναι δεδομένες για τον ρόλο που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη και ο Υπουργός Άμυνας ε, Γκέιτς τον είπα σε αυτά που είπε τοποθετήθηκε με σαφήνεια όχι για το ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν και εκείνοι δεν αναλαμβάνουν τις ε, ευθύνες τους σε σχέση με την μη αντιστοίχηση στόχων διότι γνωρίζουμε ότι και ένας από τους τελευταίους λόγους ε, του Προέδρου Μπούς ε, στο Βουκουρέστι τόνισε ιδιαίτερα ότι μια ευρωπαϊκή προσπάθεια θα πρέπει να είναι μέρος μιας διατλαντικής προσπάθειας για την ασφάλεια και την άμυνα. Μέχρι τότε όμως τα μηνύματα των Αμερικανών ήταν πολύ αντιφατικά. Και ίσως αυτό επεξηγεί γιατί δεν έκανε τη δουλειά της η Ευρώπη παρότι υπήρχαν αυτοί οι στόχοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τούτων λεχθέντων λοιπόν και ανησυχώ πραγματικά πάρα πολύ διότι πιστεύω ότι μια χώρα σαν τη δική μου η Πορτογαλία για παράδειγμα με αξιοπρόσεκτο δυναμικό δεδομένη της ιστορίας της θα χάσει αυτό το δυναμικό και αυτή θα είναι απώλεια για την Ευρώπη και για την Πορτογαλία αν δεν κάνουμε κάτι στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εν τέλει όσον αφορά τα θέματα άμυνας και το δυναμικό στην άμυνα από πλευράς μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν απευθείας. Πρώτα απ' όλα, είναι εξοργιστικό το ότι η Ευρώπη δεν καταπολέμησε τη διαφθορά στον στο πεδίο της άμυνας. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε πόρους και ένας από τους λόγους για δεν θα είναι πρόθυμοι οι πολίτες μας να υπομισθούν αυτά, αυτές τις δαπάνες στην οικονομική κρίση είναι επειδή δεν κάναμε τίποτα σε σχέση με τη διαφθορά στις ε, συμβάσεις και συνθήκες ε, για το αμυντικό υλικό και την άμυνα. Δεν είναι μόνο η διαφθορά σε σχέση με την Πορτογαλία, είναι πορτογαλική, γερμανική, αμερικανική διαφθορά. Δεν καταπολεμήσαμε λοιπόν τη διαφθορά. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε κονδύλια χρήματα σήμερα και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν θα θέλουν να δώσουν οι πολίτες τέτοια κονδύλια στην άμυνα είναι αυτός ένα σημαντικός λόγος. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκρίνατε την προσπάθειά μας στην άμυνα με τις ε, προσπάθειες των ΗΠΑ. Δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε τις προσπάθειές μας με το δυναμικό των χωρών BRICS της Βραζιλίας, Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας και να δούμε σε σχέση με το, για παράδειγμα, με την αγορά ε, από τους Κινέζους ε, δυναμικού στην Ευρώπη και τεχνολογίας. Δεν αγοράζουν οι Κινέζοι και δεν χάνουν οι Ευρωπαίοι με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις εξαγορές. Και τρίτη μου ερώτηση. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας. Η, είπατε η εκπρόσωπος ε, που δημιουργήθηκε για τις εξωτερικές σχέσεις αλλά και για τα θέματα άμυνας. Ποια διαφορά έκανε αυτή η προσπάθεια. Ανησυχήσαμε βλέποντας ότι παρόλη την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με το να πείσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, το δυναμικό τους στην Λιβύη και αυτό όχι μόνο λόγω των επιφυλάξεων κάποιων χωρών όπως της Γερμανίας, αλλά πολύ σχετίζεται αυτό με το γεγονός ότι άλλες χώρες δεν θέλουν να δαπανίσουν και να εμπλακούν σε αυτές τις δράσεις. Ποιο είδους διαφορά υπάρχει λοιπόν και ποια είναι η διαφορά που έγινε σε σχέση με τη δημιουργία του αξιώματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας για να καταφέρουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως Ευρώπη. Και εν τέλει πώς μπορούν οι αμυντικές βιομηχανίες να είναι αποτελεσματικές και να αναπτυχθούν. Γιατί αν θέλουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την ανησυχητική τάση πραγμάτων, πώς μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη και τις κυβερνήσεις ότι οι αμυντικές βιομηχανίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Γκάλ. Κύριε Γκάλ, παρακαλώ. Ähm, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τους δύο εισηγητές που ακούσαμε. Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω σε αυτό το παράδειγμα της Λιβύης και να συνεχίσω με αυτό. Ένα πολύ καλό παράδειγμα που βλέπει κανείς ότι ουσιαστικά ο ρόλος και στόχος μας θα έπρεπε να είναι τους Αμερικανούς φίλους μας που ε, δραστηριοποιήθηκαν και εν μέρη υπήρξε επιφύλαξη από πλευράς μας. Ερώτηση προς εμάς ως επιστήμονες ή για κάποιους από τους βιομηχανικούς κύκλους που παρατηρούν τα πράγματα. Πού εντοπίζετε και θέτετε εσείς τα κύρια αίτια για αυτή την επιφύλαξη που υπάρχει για μια στενότερη συνεργασία βρίσκεται πάνω-πάνω στην πολιτική ιεράρχηση των πραγμάτων στο πολιτικό επίπεδο. Είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας των στρατιωτικών μας που εκεί έχει αγκυρωθεί αυτό και έχουν μια παλαιά νοοτροπία ανεδαφική ίσως και έχουν, υπάρχουν επιφυλάξεις. Ίσως μάλλον όλα είναι οι βιομηχανικοί κύκλοι που εκάστοτε για τη χώρα τους πάντα φοβούνται και έχουν κάποιους φόβους αν υπάρχουν κάποια ανοίγματα και αν υπάρξει εντονότερη και πιο ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ χωρών ότι η οσήθιστε πορεία που ακολουθούν αυτοί οι βιομηχανικοί κύκλοι προς τα Υπουργεία Άμυνας των χωρών τους δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί και θα ακολουθηθεί μια άλλη ευρωπαϊκότερη πορεία. Ίσως πολιτικοί και στρατιωτικοί και βιομηχανικοί λόγοι που όλοι αυτοί συνδέονται και οδηγούν σε αυτές τις επιφυλάξεις. Πιστεύετε ότι μπορούμε να μάθουμε κάτι από μια ιστορία σαν τη Λιβύη υπό το πρίσμα ότι, για παράδειγμα, τι θα γίνει με την επόμενη φορά όταν θα πούν πάλι οι Αμερικανοί ότι, για παράδειγμα, δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Τι θα κάνουμε εμείς. Πιστεύετε ότι η πολιτική συζήτηση για τέτοια θέματα όταν θα έρθει η ώρα να διεξαχθεί θα προχωρήσει ή δεν έχει πολύ νόημα να στοχεύουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο. Αυτά για αυτό το θεματικό πλέγμα. Πώς αξιολογείται με άλλα λόγια και αυτό ίσως τελευταία παρέμβαση τις προσεγγίσεις ή απαρχές που υπάρχουν παρόλα αυτά στη συνεργασία μεταξύ μας. Τα παραδείγματα είναι γνωστά εξάλλου και πώς αξιολογείται τώρα αυτή την σύνθεση και συγκυρία με τους στρατιωτικούς military staff με 300 σχέδια ή προγράμματα που έχουν εντοπιστεί και όπου θα μπορούσε να υπάρξει κοινή συνεργασία. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να υπολογίζει κανείς πραγματικά ότι κάτι θα υλοποιηθεί από όλα αυτά που υπάρχουν ως προτάσεις. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το πάνελ για αυτό το pooling and sharing, αυτή την κοινή εκμετάλλευση, κοινή χρησιμοποίηση κτλ από πού βγήκε αυτή η ιδέα, η ιδέα, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ καλό για αυτούς οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν και την ευρωπαϊκή ιδέα. Μιλήσατε για αυτά τα battle groups, για αυτές τις ε, ομάδες ε, ε, μάχης κτλ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι μήπως πρόκειται για ένα σχέδιο Σούμαν που δεν, είναι, δεν έχει να κάνει τον, με τον άνθρακα αλλά έχει να κάνει με την άμυνα διότι εδώ μαζεύουμε όλες τις, όλες τις αμυντικές δυνάμεις ξηράς, αέρος, θαλάσσις, στρατιώτες κτλ. Αυτό κάνουμε. Ευχαριστώ κύριος Λίζε, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Sorry for Polish language. Συγγνώμη για τα πολωνικά. Okay. Δεν θα μιλήσω. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι σαφές ότι ακούσαμε ό,τι το καλύτερο. Για άλλη μια φορά επαναλήφθηκαν κάποια γεγονότα και δεδομένα που είναι πράγματι στοιχεία σημαντικά για την επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων και στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο υπήρξε μια διακήρυξη, μια δήλωση ενός ε, Βρετανού ναυάρχου που είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και τρεις μήνες έχει αρχίσει να χάνει το δυναμικό να χρησιμοποιεί, λέει, πυράβλους στην Λιβύη και αυτό γιατί, γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια, επαρκή κονδύλια. Και πρόκειται για μια μείωση σε μηδενικό επίπεδο. Και μάλιστα σε μια χώρα με ένα προϋπολογισμό που είναι αξιόλογος, με μεγάλες δαπάνες όσον αφορά το πεδίο της άμυνας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια τέτοια τοποθέτηση λοιπόν είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυσαναλογία μεταξύ των ε, δαπανών των Ηνωμένων Εθνών και αυτών που συμβαίνουν ε, στο αμυντικό επίπεδο από πλευρά ευρωπαϊκών κρατών με τις περικοπές. Συμφωνώ με την πλειοψηφία των παρατηρήσεων που έγιναν. Για την ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω και που είναι η εξή. Όπως βλέπετε κύριοι, η δυνατότητα να επιληθεί, να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση πρέπει να μας οδηγήσει στο να δράσουμε. Και γιατί, διότι μπορούμε να πούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια κάνοντας λόγο για τις ε, ε, αρμοδιότητες των εθνικών ε, κοινοβουλίων θα πρέπει να ε, εξοπλιστούν ώστε να μπορέσει το θέμα των ε, ε, δαπανών να προαχθεί. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα μπορέσουν να προαχθούν αυτές οι δαπάνες. Πρώτον γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια. Δεύτερον δεν υπάρχει και η βούληση να διασφαλιστούν αυτές οι δαπάνες. Δεν θα υπάρξει αύξηση λοιπόν των αμυντικών δαπανών στο πεδίο της άμυνας. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο δεύτερος εισηγητής, Μία ιδέα βλέπω να σκιαγραφείτε ότι για να εξορθολογιστούν οι δαπάνες θα πρέπει να έχουμε μια κοινή δράση σε ένα κοινό πλαίσιο. Και από τα όσα μας είπατε, μια ήπια κριτική ασκείται για το ότι έχουμε τόσα πολλά προγράμματα και σχέδια για την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρισκόμαστε στις πρώτες φάσεις και αποστέλλονται συμβολικά μηνύματα με αυτές τις δράσεις. Ερώτηση. Δεν θα έπρεπε λοιπόν τούτων όλων δεδομένων ως έχουν να εξειδικευθούμε περισσότερο, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν θα πρέπει κάποια προγράμματα να τα απαλείψουμε και να επικεντρωθούμε με τα πιο σημαντικά κονδύλια που έχουμε σε ε, πυρήνες που θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ζητεί τον λόγο. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Οι ερωτήσεις που αφορούν την επόμενη σειρά, αν θέλετε, ομιλιών, το επόμενο πάλι θα το αφήσω για αργότερα. Λοιπόν, ξεκινώντας με την κυρία Κόμες. Η διαφθορά είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Αν είναι ανάμεσα ένα, ένα θέμα από ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία δεν πάνε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Ε, το να το συνδυάζουμε με, την, ε, ε, με το θέμα της πρωτοβουλίας για την ε, ανάπτυξη της άμυνας Εάν δείτε την σημασία της αμυντικής βιομηχανίας σε σχέση με το ΑΕΠ, η ε, διαφθορά είναι αμεληταία. Η αμυντική βιομηχανία συνεισφέρει και στην, ε, συνεισφέρει στην ασφάλειά μας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Βέβαια υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και να το συνδέσω και με αυτά που είπε ο κύριος Κάλα, Δηλαδή, εάν ρωτήσετε ποιος ε, εποφελείται από την αμυντική βιομηχανία, θα έχετε και την απάντηση γιατί δεν προχωράνε τα πράγματα διότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συμμαχία, η στρατιωτική, η πολιτική, η βιομηχανία μέχρι σε έναν βαθμό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι γενικά, γενικά, και να πούμε ποιος από όλους αυτούς φταίει, θα πρέπει να δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τώρα, το θέμα της ε, Λισαβόνας και της ε, ΥΠΑ, της Αρμοστίας κτλ. Όντως θα πρέπει να ρωτήσετε την αντιπρόσωπο, την είπατε αντιπρόσωπο. Εκείνη θα πρέπει να ρωτήσετε, εκείνη θα ξέρει, εκείνη ξέρει τη δουλειά της καλύτερα. Εμείς απλώς θα παρακολουθούμε. Από το Βερολίνο. Τι μάθαμε από τη Λιβύη. Αυτό το συζητάμε γενικότερα και κάθε μέρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν να εξακολουθήσουν να μας βοηθήσουν. Δώσανε ένα, μια πρόθεση στην αρχή και μας είπαν ότι μετά θα φύγουν. Τώρα το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ηγηθεί ούτε σε ε, στρατιωτικό ούτε σε πολιτικό επίπεδο. Τριάντα χρόνια μας απασχολεί αυτό το θέμα της Ευρώπης χωρίς άμυνα. Δεν είναι για 6.000 ε, στο εξωτερικό, είναι στο, στα, 1.000, στα χίλια χιλιόμετρα. Είναι ένας δικτάτορας τρίτης κατηγορίας, αν θέλετε, την οποία δεν μπορούμε να ε, διώξουμε και δεν μπορούμε δηλαδή να προστατεύσουμε τις ε, δυνάμεις μας. Ίσως να μην έχουμε και δύναμη, τι να σας πω. Τώρα, όσον αφορά το pooling and sharing, για την Γάνδη και τα λοιπά, το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν αφήνεις αυτές τις πρωτοβουλίες στα χέρια της γραφειοκρατίας, διότι υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι συμπληρώνουν τα έντυπα και τα δελτία και υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, αν θέλετε, ε, που δεν βοηθάνε. Αυτό το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική ηγεσία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολιτική φυσιογνωμία και προσωπικό του η οποία να λέει ότι εγώ είμαι, υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία και θα την προωθήσω. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για, την, για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Εάν δεν υπάρχει κάποια πολιτική φυσιογνωμία Όπω ο, ο πρώην υπουργό άμυνα ο οποίο. Ε, ε, προσέφερε το πολιτικό του βάρος στην πρωτοβουλία της Γάνδης, δεν θα προχωρήσουν τα πράγματα. Διότι υπάρχει η γραφειοκρατία που, που μας κρατάει πίσω. Κύριε Καπέλ, το pooling and sharing δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως σας είπα, υπάρχει μια μακριά παράδοση σε αυτά τα θέματα κοινή χρήση, εκμετάλλευση κτλ. Και το Ηνωμένο Βασίλειο ξέρει πάρα πολύ καλά ε, τα θέματα αυτά έχετε 30 χρόνια ε, κοινής ε, αντιμετώπιση ε, των ενωπημένων δυνάμεων με την Ολλανδία. Και η κινητήρια δύναμη αυτή τη στιγμή που μας οθεί προς το μέλλον είναι ότι ακριβώς δεν είναι το πόσο όλοι οι στρατοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνουν ένας, αλλά υπάρχει λιβύη. Δεν μπορούμε ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη της ανικανότητας των, μεμόνων, μεμονωμένων κρατών μελών που δεν μπορούν να προσφέρουν μια ικανοποιητική άμυνα για τη χώρα του, για τις χώρες τους και τελικά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το καταφέρει αυτό. Δεν πρόκειται για σχέδιο, της, σχέδιο Σούμαν, νέο σχέδιο Σούμαν. Ούτως ή άλλως η, πολιτική άμυνας και ασφάλισης δεν είναι η κινητήρια δύναμη που θα ενοποιήσει την, την Ευρώπη. Αυτό το έχουμε ε, δει και στο παρελθόν δεν χρειάζεται να τρέχουμε ψευδεστήσεις. Κύριε Λίζεκ, ούτως ή άλλως το θέμα δεν είναι η εξειδίκευση η οποία τώρα γίνεται, γιατί όλοι εξειδικεύονται στο φθηνότερο, είναι θέμα συντονισμού. Θα πρέπει να μιλάμε όλοι ο ένας τον άλλον. Μέχρι και σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας δεν μιλάνε μεταξύ τους. Είναι αστείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχετε δίκιο κυρία Γκόμες το να κάνουμε τις συγκρίσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν είναι σωστό διότι είναι διαφορετική κλίμακα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ευρωπαϊκές ε, αμυντικές δαπάνες με τις αμερικανικές διότι μιλάμε για κρατικές, για εθνικές άμυνες. Ίσως έπρεπε επομένως να διαρρέσουμε δια του 27. Επομένως, η σύγκριση με άλλες χώρες θα ήταν ε, ε, χρήσιμο εάν συγκρίνουμε ας πούμε την Γαλλία και τη Γερμανία όσον αφορά τις, ε, τις δαπάνες αλλά όχι να τις συγκρίνουμε αυτές τις χώρες με, την, με την, τις Ηνωμένες με το Ισραήλ την Κορέα ενδεχόμενα Πολλές ερωτήσεις έγιναν για τις δυνατότητες συντονισμού των προσπαθειών γίνεται η οικονομική εδώ ανάλυση της θεωρίας των συμμαχιών. Η συμμαχία, η συμμαχία, το ΝΑΤΟ είναι το καλύτερο παράδειγμα. Εάν δούμε ότι η κοινή χρησιμοποίηση των μέσων τελικά είναι αμελητία σε σχέση με τον προϋπολογισμό, διότι το 1% των δαπανών ε, χρησιμοποιείται από κοινού. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωράει. Ίσως θα έπρεπε να δούμε πώς η θεωρία των συμμαχιών θα μπορούσε να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εδώ όμως είναι ένα θέμα ομοσπονδίας αν θέλετε. Εδώ δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να συνεργαστεί κανείς ή να προσφέρει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και δεν υπάρχει και κάποιος περιορισμός. Ε, όμως εάν δούμε τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο αν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πιέζει αν θέλετε ε, τους εταίρους οι εταίροι δεν κάνουν τίποτα. Τώρα, για τις ε, συνέπειες ε, που θα είχε μία απόφαση των Υπουργών στα θέματα ανάπτυξης. Να σας να επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως για τις ε, συνέπειες κλίμακας, για τα αποτελέσματα κλίμακας. Δύο Ισραηλινοί επιστήμονες έχουν πει, έχουν αποδείξει ότι το να δαπανούμε λίγα ή τίποτα είναι το ίδιο πράγμα. Επομένως, εάν η είσοδος, αν θέλετε, είναι υψηλή, ε, κοστίζει πολύ δηλαδή, δεν θα μας ακολουθήσουν μετά. Δεν θα υπάρχει επένδυση σε όσον αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία. Τώρα, το πρόβλημα είναι η βιομηχανία άμυνας ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που έχει και σε μη στρατιωτικό επίπεδο. Βλέπουμε ποιος, ποιος είναι ο μηχανισμός εδώ ε, και ο μηχανισμός αυτός περιορίζεται βέβαια διότι είναι και περιορισμένη σε η βιομηχανία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και Κάμπελ για τον Ευρωπαϊκό στρατό. Θα ήταν ίσως το ιδανικό αυτό, αλλά ε, τα θέματα των αποστολών και των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέτει ένα θέμα ομοσπονδίας, διότι εδώ θα πρέπει να, μπορούμε, να καλύψουμε και τις μη προβλεπόμενες δαπάνες που θα μας επέτρεπαν αυτές οι επιχειρήσεις να γίνουν κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Όμως, εάν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό project, ούτως ή άλλως οι δαπάνες και επομένως και οι προσπάθειες ε, είναι κατανεμημένες. Κύριε Λίζεκ, το θέμα το οποίο τίθεται είναι θέμα πολιτικής φιλοδοξίας. Ούτως ή άλλως οι προσπάθειες άμυνας είναι θέμα πολιτική πολιτικής βιομηχανίας. Ο καθηγητής και στο ΜΑΙΤΙ μας είπαν ότι το 5% των, ε, του αμερικανικού προπολογισμού είναι ε, ε, για την άμυνα. Στην Ευρώπη το 2% δεν είναι. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Μου είπε, μου έλεγε ότι στο πόλεμο της Κορέας οι Αμερικανοί ε, δαπανούσαν το 10% και αυτό από την κοινωνία τους πολίτες ήταν αποδεκτό. Εδώ είναι θέμα και στην Ευρώπη, είναι θέμα πολιτικής απόφασης, ε, είναι θέμα πολιτικού οράματος. Τώρα, όσον αφορά για την βιομηχανία άμυνα ή τον προπολογισμό άμυνα είτε για αποστολέ, ε, δεν, είναι το θέμα, δεν πρέπει να βλέπουμε το θέμα καθαρά από οικονομικούς όρους. Είναι θέμα πολιτικής φιλοδοξίας και από εκεί και πέρα για τον τρόπο που θα γίνεται η κατανομή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν μπορεί όλοι να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα θα έχει πει αυτά. Ε, δεν μπορεί όλοι να κάνουμε την, την ίδια δραστηριότητα. Από οικονομικής πλευράς αυτό είναι άσκοπο. Βέβαια η βιομηχανία προσπαθεί να ε, προστατεύσει τις αγορές, ε, το κεκτημένο, αλλά το πρόβλημα είναι να δούμε και πόσο συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη. Εάν ε, δούμε πόσο διαχειριζόμαστε τα προγράμματα συνεργασίας, αυτά τα προγράμματα δεν είναι τελικά αποτελεσματικά. Αλλά δεν φταίει το πρόγραμμα αυτό, αυτό καθεαυτό, φταίει ο τρόπος διαχείρισης που εξαρτάται από τις εθνικές ε, αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις ε, οικονομίες κλίμακας που θα μπορούσαμε να κάνουμε, παραδείγματο χάρη για την κατασκευή ε, αεροσκαφών ή για την κατασκευή κάποιων δυνατοτήτων, κάποιο μέσον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για το δεύτερο πανελ έχω την χαρά να καλωσορίσω τον εταίρο του Βασιλικού Ιδρύματος ε, για τις ε, στρατιωτικές ε, ικανότητες τον κύριο Τόμας Χέσεκ και επικεφαλής του κέντρου στο Λονδίνο και τον κύριο Γκραμ ε, Uh, Έχουμε τις προοπτικές ε, για τις συμπράξεις ε, και τις κοινέ δράσεις, ιδιαίτερα για το ποιο στρατιωτικό δυναμικό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για αυτές τις συμπράξεις και ποιες είναι οι κύριες πολιτικές δυσχέρειες που μπορεί να συνδέονται με αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την δυνατότητα ε, διασυνδεσιμότητας και λειτουργικότητας. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε πράγματι ευκαιρίες ε, για τη σύμπραξη και κοινέ δράσεις. Θα ήθελα να σας εκθέσω έξι ιδέες ε, για αυτά τα θέματα απόψε παραμένοντας μέσα στο πλαίσιο των ε, αρμοδιοτήτων μου. Πρώτο στοιχείο, η σύμπραξη και οι κοινέ δράσεις δεν είναι τίποτα καινούριο και έχουμε μια μακρά ιστορία που έχει 60 χρόνια ήδη ε, δραστηριότητες στη σύμπραξη και κοινέ δράσεις. Κάνοντας λόγο για αυτή τη σύμπραξη και τις κοινέ δράσεις, η έμφαση είναι πάντα στην περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, σε σχέση με την περιφερειακή συνεργασία, έχει τις αξίες της και πρέπει να δούμε και ποιες είναι αυτές οι, αυτά τα θετικά. Όμως, σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες που μπορούν να δώσουν νέα προγράμματα στην περιφερειακή αυτή σύμπραξη και ανάπτυξη ή να αναβαθμίσουμε το επίπεδο αυτής της περιφερειακής συνεργασίας σήμερα. Όμως η ιδέα δεν είναι να κατακαιρματιστεί η Ευρώπη σε νησίδες περιφερειακής συνεργασίας. Πρέπει να προσβλέψουμε σε ένα είδος δικτύου, διευρωπαϊκού δικτύου, διευρωπαϊκών συνεργασιών και γι' αυτό από την δική μου πείρα πρέπει να πω ναι στην περιφερειακή συνεργασία. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε τη σύμπραξη και τις κοινέ δράσεις σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμπραξη και κοινέ δράσεις για ένα συγκεκριμένο κοινό σύστημα εξοπλισμών έτσι μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα win-win, θετικό για αμφότερες ε, τις πλευρές. Και η δυνατότητα αύξησης του δυναμικού είναι μεγαλύτερη και επιπλέον έχουμε δυναμικό το οποίο παρέχεται για να μπορέσουν πολλές χώρες να συμμετάσχουν μεγαλύτερες και μικρότερες πανευρωπαϊκά σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη ιδέα λοιπόν. Είναι περιφερειακή αυτή η συνεργασία βέβαια όμως επίσης υπάρχει η σύμπραξη και κοινέ δράσεις σε εξειδικευμένους τομείς και συγκεκριμένες προτεραιότητες. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι ότι πολύ συχνά όταν κάνουμε λόγο για κοινέ δράσεις και σύμπραξη πολλές φορές πιστεύει κανείς ότι συγκρίνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα μια χώρας. Το αντίθετο συμβαίνει και θα το αποδείξω για παράδειγμα στην Ολλανδία, στη χώρα μου. Έχουμε θεσπίσει κοινά, ε, κοινό επιτελείο όσον αφορά τη σύμπραξη και τις δράσεις. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι αν κάτι τέτοιο θεωρείτε ότι πάει υπερβολικά μακριά, παρόλα αυτά μπορεί να συμπράξει μια χώρα χωρίς να απολέσει καθόλου τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στα διάφορα δορυφορικά προγράμματα που έχουμε στην Ευρώπη. Η χώρα μου, το Βέλγιο και συμμετέχουν και άλλοι έχουμε 6 έως 10% των, ε, του συνολικού κόστους και σαν αποτέλεσμα η χώρα μου έχει την δυνατότητα να επανακατευθύνει δορυφόρους και να ζητήσει να δοθούν συγκεκριμένες εικόνες πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, time slot. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και είναι στα χέρια μας και αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο συνδέεται σε σχέση με το ποσοστό δικής μας σύμπραξης θα έλεγα μεγάλης ε, αποδοτικότητας. Ε, διαφορετικά δεν θα υπήρχε μια τέτοια αποδοτικότητα. Στο τέλος τέλος λοιπόν τα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει κανείς είναι να ασκήσει επιρροή στην λήψη αποφάσεων όσον αφορά άλλους και να επιτύχει αποτελέσματα επηρεάζοντας ε, τις αποφάσεις. Η σύμπραξη και οι κοινέ δράσεις είναι ακριβώς ένα μέσο για να πετύχουμε αυτό εξαρτάται από το πώς θα διοργανώσει κανεί τη σύμπραξη και τις κοινέ δράσεις. Τρίτη παρατήρηση. Έχουν τα όρια τους οι συμπράξεις και οι κοινέ δράσεις, διότι σε ένα κοινό καλάθι εντάσσουμε αυτά τα οποία ήδη υφίστανται και υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας. Το 2001 εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> εντοπίσαμε ποιε ήταν οι απαιτήσει και ταυτόχρονα εντοπίσαμε και ποιες ήταν και οι ελλείψεις ή τα κενά σε στρατηγικό επίπεδο. Παρόλε λοιπόν τις συμπράξεις και κοινέ δράσεις που υπήρξαν από το 2001 μέχρι σήμερα, 2011, οι στρατηγικές ελλείψεις εξακολουθούν να υφίστανται αναλύωτες. Έχουμε τα πέντε διαρκεί μόνιμα χαρακτηριστικά των ε, δυνατοτήτων της Ευρώπης. Περισσότεροι ε, στρατιώτες, γυναίκες και άνδρες σε σχέση με τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τις κοινέ δαπάνες των 27 κρατών μελών, <clears throat> σε παγκόσμιο επίπεδο δεύτεροι είμαστε. Τρίτο χαρακτηριστικό, στο επίπεδο των 27 κρατών μελών έχουμε πολλές συγκεκριμένες ε, δυνατότητες στρατιωτικές που πλεονάζουν, είναι πλεονασματικές. Αντίθετα, έχουμε πολλές ε, ελλείψεις στο στρατηγικό επίπεδο, αναλύωτα. Παρ' όλα αυτά, είμαι αισιόδοξο, διότι υπάρχει ένα πέμπτο χαρακτηριστικό στοιχείο και είναι πολύ ενδιαφέρον να το σημειώσει κανεί αυτό τα πλεονάσματά μας αντισταθμίζουν τις ελλείψεις μας και αυτό είναι σημαντικό. Το μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα να αποστείλω είναι ότι οι συμπράξεις και οι κοινέ δράσεις που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε και έχουμε στα χέρια μας σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα, για ένα ευρύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα, για πιο μόνιμα χαρακτηριστικά διαρθρωμένης, δομημένης συνεργασίας και σχεδιασμού, προγραμματισμού στο αμυντικό επίπεδο, στοχεύοντας και προσανατολιζόμενοι πάντα στο να καλύψουμε τις στρατηγικές μας ελλείψεις και τα κενά και ίσως ε, με μια πιο δομημένη, διαθρωμένη τέτοια και πιο σταθερού χαρακτήρα, μόνιμου χαρακτήρα συνεργασία, ένα από τα κριτήρια αυτής θα πρέπει να είναι να διατηρήσει και ή δυνατόν να αυξήσει κιόλας ε, τα δικαιώματα των συμμετεχόντων όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Οι συμπράξεις ε, και οι κοινέ δράσεις είναι λοιπόν ένα πρώτο, μια πρώτη φάση. Πρέπει εδώ να ε, κάνουμε μια παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ υψηλέ προσδοκίες για τις συμπράξεις και τις κοινέ δράσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πνεύμα της Γάνδης θα παραμείνει ζωντανό και θα συνεχίσει να δρά. Και έτσι λοιπόν η σύμπραξη και οι κοινέ δράσεις δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα καταχρώμεθα και θα πρέπει να εποφελούμεθα όλοι και σε σχέση με τη συνέχιση των ε, μέχρι σήμερα δράσεών μας θα μπορούσε κανείς ε, σε επουσιοδέστερα σημεία να επικεντρώνεται και ε, να συνεχίσει να δρά Έχουμε κάποιες ε, ενδείξεις ότι προς αυτή την κατεύθυνση κάποιοι κινούνται. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα της Γάνδης ζωντανό και να διασφαλίσουμε ότι το πρώτο βήμα το οποίο εκπονούμε τώρα θα είναι σημαντικό γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν είναι σημαντικό αυτό το πρώτο βήμα, δεν θα υπάρξει δεύτερο βήμα και δεν θα υπάρξει ένας πιο διαθρωμένος, ε, μια πιο διαθρωμένη και δομημένη προσέγγιση και θα αποβιώσει αυτή η ε, πρωτοβουλία, δεν θα έχει μέλλον με άλλα λόγια. Αυτό είναι λοιπόν κρούχοδονα κινδύνου να το λάβουμε υπόψη. Συμπράξεις και κοινέ δράσεις. Να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να αναζητήσουμε εκείνα τα προγράμματα και σχέδια που συνενώνουν χώρες και τις συνδυάζουν με τέτοιο τρόπο σε θελούσια βάση εθελοντικά ώστε να έχει επίπτωση στο σχεδιασμό του στον αμυντικό με θετικό πνεύμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με την Ολλανδία και το Βέλγιο <clears throat> παρόλα τους ε, τα κυριαρχικά δικαιώματα κανείς στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία δεν θα αναπτύξει προγράμματα και σχέδια που να αφορούν τον εξοπλισμό του ναυτικού χωρίς να υπάρχει διαβούλευση της άλλης χώρας. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχει επίπτωση και στο σχεδιασμό των αμυντικών δράσεων αμφωτέρων των χωρών με θελοντική θελούσια βάση αλλά με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ δράσεις και συμπράξεις. Λοιπόν, ένα πρώτο βήμα είναι αυτό και πρέπει να είναι ένα σημαντικό ζωοποιό πρώτο βήμα. Εύκολο να το πει κανεί αυτό βέβαια. Μπορούμε να, να το κάνουμε. Έχουμε παραδείγματα για κάτι τέτοιο. Για μένα ήταν εύκολο να βρω κάποια τέτοια στοιχεία διότι απαριθμούνται σε, μια μελέτη που υιοθετήθηκε στις 11 Μαΐου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο πρωτοβουλίες βρισκόντουσαν εκεί. Η δημιουργία ενός κέντρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε δράσεις πρόνοιας και πρόληψης να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται συνενώνοντας όλες ε, τις εμπλεκόμενες δυνάμεις ε, για την διαχείριση κρίσεων και σειράξεων. Και ένα δεύτερο παράδειγμα για την ε, βελτιωμένη αντιμετώπιση αυτών των αμυντικών σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, αν υλοποιηθεί αυτό, τα κράτη-μέλη θα έχουν ένα σαφέστατο μήνυμα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συμπράξεις και κοινέ δράσεις στον αμυντικό τομέα. Και το δεύτερο, με κοινό επιτελείο, είναι μια πραγματιστική λύση με βάση τα μαθήματα που έχουμε συναγάγει και θα δημιουργήσει μια κερδοφόρα κατάσταση όχι μόνο για τα θεσμικά οργάνα αλλά και για τα κράτη-μέλη κατά πρώτο λόγο. Και η παρατήρηση Έκτη παρατήρηση. Όλα αυτά είναι εφικτά, μπορούν να υλοποιηθούν. Νομίζω ναι. Πρώτα απ' όλα έχουμε την, ε, το πρόγραμμα λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όμως πρέπει να το πούμε αυτό θα έπρεπε να μπορέσει να, να διασφαλιστεί ότι θα βοηθηθεί αυτό το πρόγραμμα με κάθε τρόπο. Δεύτερον, να επηρεάσουμε τους πολίτες, την κοινή γνώμη. Και συνολικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες μας είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ μιας Ευρώπης που θα είναι σε θέση να κάνει κάτι το σημαντικό για λογαριασμό της. Έχουν όμως και κριτικές παρατηρήσεις οι πολίτες μας ταυτόχρονα και υπάρχουν λόγοι για αυτές τις κριτικές παρατηρήσεις. Είχαμε το πρόβλημα του πόλεμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, το δεύτερο, τον πόλεμο στον στο Ιράκ, το τρίτο προηγούμενο είναι η σημερινή περίπτωση του πολέμου στη Λιβύη. Είναι τρεις φορές που έχουν παρουσιαστεί τέτοια προβλήματα και πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούμε. Και επιπλέον πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και σταράτα. Για άλλη μια φορά προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες το μήνυμα. Και τώρα είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να δράσετε αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνετε κάτι ώστε να είσαστε αποτελεσματικοί με το στρατιωτικό δυναμικό σας. Δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια και ποτέ δεν υπήρχε και τώρα είναι σαφές για όλους ότι δεν υπάρχει πλέον ανταγωνισμός σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το αντίθετο. Και αυτό που βλέπουμε είναι τέλος ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει μια αυξητική τάση να αφήνονται ε, θέματα που αφορούν το στρατηγικό επίπεδο, τη, τη στρατηγική συνιστόσα, να μην αφήνονται αυτά στο εθνικό επίπεδο και γίνεται η προσπάθεια να ενταχθούν σε ένα υψηλότερο, ε, σφαιρικότερο επίπεδο. Είμαι και αισιόδοξο όμως γιατί υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να δράσουμε στρατηγικά ενωμένοι και με συνεργασία ιδιαίτερα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βουλευτές που επιτροπή σας ευχαριστώ πολύ που δώσετε το λόγο. Θα σας μιλήσω για την πολιτική του pooling και sharing και ίσως απαντήσω στα ερωτήματα Γκάλερ και Λίσεκ πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να ε, έχουν μεγαλύτερη ε, συμμετοχή σε αυτές τις κοινέ προσπάθειες και ίσως και ασχοληθώ με αυτά που είπε και η κυρία Γκόμε. Surviving Austerity είναι μια μελέτη που διασημοσιεύτηκε τον Μάιο και μου ζήτησαν πριν από ένα χρόνο να δω παραδείγματα του παρελθόντος, ε, αν υπήρξαν επιτυχίες ε, και πού υπήρξαν αποτυχίες, στο pooling και sharing. Η λογική είναι απλή. Ε, είναι, έχει άμεσο οικονομικό νόημα αυτή η κοινή εκμετάλλευση. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έχουν ακουστεί και υποθεί πολλά, αλλά δεν έχει ε, συνοδευτεί όλη η προσπάθεια από την ανάλογη επιτυχία. Οι δημόσιες συμβάσεις, ναι, αλλά σε ό,τι αφορά τις δομικές ε, κοινέ δομικέ μονάδε, παραδείγματο χάρη, τι κοινέ υποδομέ, αυτό είναι κάτι σπάνιο. Από τα 1,6 εκατομμύρια ένστολου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο λίγε χιλιάδε είναι σε μόνιμα ενοποιημένε ε, μονάδε. Και το 90% περίπου των ε, εξοπλισμών είναι εθνική και όχι ευρωπαϊκή. Τα μέλη της ε, υποεπιτροπής είστε πολιτική, αντιμετωπίζεται πολιτικά εμπόδια αυτή της ολοκλήρωσης. Οι χώρες όμως πιστεύουν ότι αν έχουν μονάδες τους, οι δυνάμεις τους σε άλλες χώρες μπορεί να αναγκαστούν να πολεμήσουν πολέμους που δεν τους επιθυμούν. Αλλά θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις. Ε, άλλες ε, χώρες ανησυχούν επίσης για την εγκατάλειψη. Δηλαδή αν είναι σε μια κοινή ε, ομάδα, σε μια κοινή δύναμη, μπορεί να μην τους δοθεί δυνατότητα όταν χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν μια ομάδα μάχη, με παραδείγματος χάρη. Και επίσης υπάρχει και η περίπτωση κάποιοι να χρειαστεί να προσπαθήσουν να επιτύχουν στόχους άλλων χωρών. Ο ταξίαρχος μας μίλησε για κάποια παραδείγματα επιτυχίας, ε, το βελγολανδικό παράδειγμα ή ένα άλλο παράδειγμα, ε, η αμφίβια μονάδα. Γιατί λοιπόν κάποιες ιστορίες στέφονται με επιτυχία και κάποιες όχι. Υπήρξαν ε, κάποια αμυντικοί σύμβουλοι, υπουργοί κτλ. οι οποίοι συζήτησαν πρόσφατα για τους παρελθούσες εμπειρίες τους και εντόπισαν κάποια βασικά διδάγματα τι κάνει η επιτυχία στο pooling and sharing. Δεν θέλω να σας εκθέσω όλα τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία περιλαμβάνονται και στη μελέτη, αλλά σε πέντε θα επικεντρωθώ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι Αυτές οι πέντε παρατηρήσεις φυσικά δεν είναι γραμμένες σε μάρμαρο και φυσικά θα πρέπει να δοκιμαστούν κατά πόσο θα βοηθήσουν να επιτύχει γενικότερα το pooling and sharing. Πάντως είναι πέντε επιτυχημένες ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Είναι να βρει κανείς έναν εταίρο που θα έχει παρόμοια στάση, παρόμοια στρατηγική κουλτούρα και προθυμία. Να είναι είτε παγκόσμιος είτε τοπικός παίκτη. Σε διαφορετική περίπτωση, ε, το είδαμε αυτό, ε, η γερμανική ταξιαρχία στο Αφγανιστάν δεν λειτουργήσε. Γιατί υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί και έτσι και ιδίω το ε, Γερμανικό Υπουργείο Άμυνα ε, είναι πάρα πολύ απρόθυμο να κάνει κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον. Τα μα τα είπε και ο Δόκτωρ ε, Μέλινγκ. Σε άλλε περιπτώσει λένε ότι πρέπει να είναι κοινέ οι αντιλήψει με τον εταίρο ή να υπάρχει η ίδια προθυμία, η ίδια δυνατότητα να είναι κάποιος ένας παγκόσμιος στρατιωτικός εταίρος. Και μπορεί κάθε χώρα να επιλέξει πού θα επικεντρωθεί σε ποια ε, κατεύθυνση, όπως παραδείγματος χάρη υποδομές. Και αυτό φαίνεται να επιλέγει η Γερμανία προς το παρόν. Επίσης πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, είναι ένα άλλο συστατικό επιτυχίας ένα ε, δίδαγμα πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω όταν κάποιος ε, θα προχωρήσει σε συμπράξεις για την αυτοάμυνα. Θέλουμε τότε να είμαστε σίγουροι ότι ο ατέρος που επιλέξαμε δεν θα μας αναγκάσει να μην χρησιμοποιήσουμε για την αυτοάμυνά μας κάποιες δυνάμεις. Ε, γι' αυτό οι βόρειες χώρες Τους αρέσει πάρα πολύ να ακολουθήσουν αυτή την ε, προσέγγιση για την ασφάλεια του ανώτατου βορρά. Είναι η αυτοάμυνα κάτι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τρίτη παρατήρηση. Οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να είναι σε ισότιμο επίπεδο ανταγωνιστή ό,τι αφορά τις αμυντικές εταιρείε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα εξοικονομεί κανείς πόρους γιατί έχει λιγότερες ε, υποδομές αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια εταιρεία εκεί έξω, η οποία θα είχε πάρει μια σύμβαση που δεν θα την πάρει με αυτή την περίπτωση. Για να αποδώσει λοιπόν το pooling and sharing θα πρέπει να υπάρχει μια ισοτιμή, ισομερή κατανομή αυτών των απολειών. Για τη διαφορετική περίπτωση θα δει κανεί, ε, παραδείγματο χάρη έγινε με την Βρετανία, που κάποιοι με τη Γαλλική Συμφωνία δεν έχουν ε, ικανοποιηθεί γιατί θεωρούν ότι θα χάσει η ε, αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή υπάρχει μεγαλύτερο προστατευτισμός στην Γαλλία και ίσως μάλιστα αρθεί και η στήριξη ε, για τη συνθήκη αυτή αν μάλιστα αυτό θα γίνει από τη γαλλική πλευρά αν χάσουν ε, οι εταιρείε ε, τι συμβάσει του. Επίση, σαφεί προθέσει είναι ανάλυση συστατικό επιτυχία, πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριο Κάμπελ μίλησε για του διάφορου λόγου που μπορεί να οδηγήσουν σε χώρε αυτή την σύμπραξη, την κοινή εκμετάλλευση. Παραδείγματο χάρη, Ευρωπαϊκό στρατό, η εξοικονόμηση πόρων, η να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης, ε, η, η Τουρκία κτλ. Εξομάλυνση διαφωνιών ε, μεταξύ χωρών που δεν ήταν φιλιρινικές μεταξύ τους. Πάντως πάντοτε θα επικεντρώνεται κανείς σε μια κοινή, χάρη, κοινή ταξιαρχία για έναν ευρωπαϊκό στρατό ή συνένωση εκμετευτικών εγκαταστάσεων και ευκολιών αν θέλει κανείς να εξοικονομήσει πόρους. Πάντως πρέπει να είναι σαφείς οι προθέσεις γιατί γίνεται το κάθε τι. Έτσι αποφεύγονται δυσκολίες όταν θα πρέπει να επιλεγεί η δυνατότητα η συγκεκριμένη. Πέμπτη παρατήρηση και τελευταία. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Η κυρία Γκόμες το είπε. Πράγματι, η διαφθορά είναι πρόβλημα. Όταν δημιουργούν μονάδε οι κυβερνήσει, θέλουν να εξορθολογήσουν ίσω και να συγχωνεύσουν τι διαδικασίε ε, διαγωνισμών του. Αυτό σημαίνει όμω ότι κάποιοι εθνικοί υπάλληλοι θα αναγκαστούν να μοιραστούν ε, ή ίσω και να χωρίσουν τελώ τι δυνατότητε και τι εξουσίε ε, λήψη αποφάσεων. Αν υπάρχει κάποιο διεφθαρμένο υπάλληλο, αυτό θα θεωρήσει ότι απειλείται από το pooling και εσέν. Και αν μπορεί να επηρεάσει επαρκώ την κυβέρνηση, ίσω ε, θα μπορούσε και να το υπονομεύσει το pooling και sharing. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα έχω αντλήσει από τις παρελθούσες εμπειρίες pooling και sharing. Δεν θέλω να σας κουράσω, έχω πάρα πολλά παραδείγματα στο έγγραφο που έχω εκπονήσει και θα ήθελα τώρα να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Τι μπορούμε να αντλήσουμε ως δίδαγμα για το μέλλον. Και μετά θα κάνω και κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής. Το σημαντικότερο συμπέρασμα για τη μελλοντική πολιτική είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει να υπάρξουν πολλοί παράγοντες για να επιτύχει το pooling και sharing. Αλλιώς θα είναι εξαίρεση και όχι κανόνα σε κοινέ μονάδες. Ή μπορεί να είναι επιτυχημένα παραδείγματα μόνο σε κάποιες χώρες ε, που μπορεί να μην είναι κοντά γεωγραφικά μόνο, αλλά να έχουν παρόμοια στάση απέναντι στη βιομηχανία, παρόμοια στρατηγική νοοτροπία ή πόψεις για την άμυνα, παρόμοια στάση για την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη κτλ. Αλλά μάλλον δεν θα βρει κανεί εύκολα πολλέ χώρε που θα πληρούν αυτέ τι προποθέσει πέραν τη στενότερη γεωγραφική περιοχή. Καλό είναι πάντως να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία πολλαπλών συμβατών εισίδων συνεργασία. Συμφωνώ με τον ταξιάρχο ε, στα πιο πολλά, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο ε, διαφωνώ. Βέβαια, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ, διαφορούμε σε κάποια σημεία και μπορούμε να τα συζητήσουμε εδώ ίσως. Αυτές είναι οι σύνδες ε, περιφερειακές ήδη υπάρχουν. Έχουμε τη Γαλλία και την Βρετανία. Έχουμε τις χώρες του Μπενελούξ βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, Τσέχ και Σλοβάκη επίσης. Ε, μεγαλύτερη συνεργασία, από των και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης θα μπορούσαν να συγκροτήσουν σύντομα μια τέτοια νησίδα συνεργασίας. Αλλά ε, επειδή θα πρέπει να να υπάρξει ευθυγράμμιση πολλών παραγόντων, νομίζω ότι το pooling και sharing καλύτερα γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Δεύτερον, τι είδου δυνατοτήτων αυτέ οι νησίδε θα πρέπει να επιλέξουν να συνενώσουν και να χρησιμοποιήσουν από κοινού και με ποιον. Αν οι κυβερνήσει επικεντρωθούν ε, στην ολοκλήρωση μη αναπτύξιμων, μη μάχημων ε, δυνάμεων, θα θέλουν να τι χρησιμοποιήσουν. Ε, ίσως θα είναι πιο εύκολο σε σχέση και με το γαλλογερμανικό παράδειγμα. Είδαμε αν υπάρχουν ασύμβατες στρατιωτικές νοοτροπίες Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξη μια μονάδα, αλλά ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται ποτέ αυτή η δυνατότητα. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτέ οι μονάδε για τη συντήρηση ή για άλλε υποδομέ. Επομένω, δεν θα σταλούν ποτέ στο πεδίο τη μάχη. Για το μέλλον, ένα άλλο δίδαγμα. Τα εμπόδια στην ολοκλήρωση είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτέ οι συνεισίδε συνεργασία είναι διαφορετικέ η μια από την άλλη και οι περιφερειακές αυτές διαφορέ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να έχουμε προσαρμοσμένε ανά γεωγραφικό τμήμα στρατηγικέ. Οι Γερμανοί είπαμε ότι είχαν κακή εμπειρία με την ανάπτυξη δυνάμεων, άρα στην περίπτωσή του θα πρέπει να ολοκληρώνουν, να συνενώνουν μη μάχημε ομάδε. Η Γαλλία, η Βρετανία θα πρέπει να εφαρμόσουν την συνθήκη την οποία έχουν υπογράψει. Θα μπορούσαν, όπω είπαμε, να έχουν μια συνεργασία των αμυντικών του δυνάμεων, όπω έχει γίνει από τον πυραυλικό τομέα. Η Τσεχία και η Σλοβακία που έχουν συνομιλίε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνήσουν τους τομείς συνεργασίας που είναι πλέον ελπιδοφόροι και έχουν το λιγότερο πολιτικό κόστος. Και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ήδη εταιρική σχέση, έχουμε την σκανδιναβική συνεργασία, θα πρέπει να δουν σας περισσότερο τη δομική ε, διάσταση. Και ίσως καταλήξουν και στη δημιουργία κοινών μονάδων. Επίση, οι κυβέρνησε δεν θα πρέπει να δημιουργούν ταυτόσιμου ομίλου, ταυτόσιμε ομάδε. Κάθε νησίδα θα πρέπει να είναι διαφορετική, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ ανάγκε, διαφορετικέ χώρε και διαφορετικοί προπολογισμοί. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί ίσω θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο επίπεδο αυτάρκεια και θα μπορούσαν να αναπτύσσουν και μεγάλες εθνικές δυνάμεις στις διάφορες αποστολές. Οι μικρομεσαίες χώρες μάλλον θα πρέπει να, είναι πιο, ε, να έχουν πιο ισχυρέ σχέσεις αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης για μεγαλύτερη ολοκλήρωση και δεν έχουν πολλές επιλογές. Ορισμένα μικρομεσαία κράτη ίσως χάσουν εάν δεν ε, μοιραστούν τις δυνατότητές τους γιατί δεν έχουν τους πόρους να χρηματοδοτήσουν τα σχετικά και ολοκληρώνοντα με αυτά τα διδάγματα και μετά θα περάσω σε κάποιε συστάσει, νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το pooling και sharing θα πρέπει να περιλαμβάνει, να έχει τη συμμετοχή και τη βιομηχανία αυτή εξ αρχή. Γιατί αν μείνουν εκτό των διαβουλεύσεων οι εταιρείε, δεν θα μπορούν να ε, μιλήσουν για τι επιπτώσει που έχει το pooling και sharing και ίσω μάλιστα να ασκήσουν πιέσει κατά τη συνεργασία. Φοβούμαι ότι θα χάσουν ε, την ε, επιχειρηματική του δραστηριότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει από την αρχή να συμμετέχουν σε συνομιλίε οι εταιρείε και να στηρίζονται οι συγχωνεύσει των εταιριών ώστε να είναι ε, πιο εύκολη η δημιουργία μια σταθερή βιομηχανική βάση. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, κάποιε συγκεκριμένε συστάσει πολιτική. Φαντάζομαι διαπιστώσατε ότι στην παρουσίασή μου τονίζω τα κράτη-μέλη και δεν μιλώ τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένο οι κυβερνήσει παραμένουν αποφασισμένε να προασπιστούν την κυριαρχία του, την εθνική κυριαρχία του στα στρατιωτικά θέματα. Και αυτό θα ισχύσει και τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν πολύ χρήσιμα πράγματα που μπορεί άμεσα να κάνει σήμερα μέσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερι διαφορετικέ κατηγορίε, αλλαγή νοοτροπία, δημιουργία κινήτρων, απομάκρυνση εμποδίων, διαχείριση δυνατοτήτων. Πρώτον, με τι νοοτροπίε εδώ το βασικό εμπόδιο είναι η άγνοια. Το pooling και sharing είναι σαν την παγκόσμια ειρήνη. Όλοι θέλουν, όλοι είναι υπέρ, αλλά κανεί δεν ξέρει πώ να το πετύχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν πρωτοβουλίε περιφερικέ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, ε, συστηματική συλλογή δεδομένων ε, σε σχέση με την επιτυχία και την αποτυχία κάποιων παρελθόντων προγραμμάτων για να λυθούν διδάγματα και νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την εκπόνηση των μελλοντικών στρατηγικών που μετά θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα πολύ σημαντικό ε, εργαλείο που έχει Ένωση είναι ε, αυτό το κολέγιο της άμυνας και ασφάλειας. Επίσης έχουμε τις μάχημες ομάδες, τα battle groups που όταν ε, δημιουργήθηκαν ήθελαν να ενθαρρύνουν την μόνιμη συνεργασία ίσως και την ολοκλήρωση που δεν έγινε όμως γιατί αυτό γίνεται εκ περιτροπής για έξι μήνες και μετά πάλι χωρίζουν οι δρόμοι των κρατών. Νομίζω ότι η Πολωνία θα πρέπει αυτά τα battle groups να έχουν μια εκ περιτροπής ε, διάσταση τρία χρόνια ίσως, αλλά να είναι οι ίδιοι εταίροι. Δηλαδή πάντοτε η Πολωνία με τις χώρες Βαλτικής ανά τρία χρόνια και έτσι μπορεί να υπάρχει αυτή η μόνιμη συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Έχει γίνει και κατά το παρελθόν τέταρτη σύσταση την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για την άρση των εμποδίων. η το κάνει μάλιστα, μάλιστα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την οδηγία για τους ε, διαγωνισμούς ε, για αμυντικούς εξοπλισμούς. Ήδη γίνεται ε, μείωση φραγμών για το διασυνοριακό εμπόριο. Αυτό μπορεί να συζητηθεί παραδείγματος χάρη με εναρμόνιση των τάσεων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και αποθάρρυνση των χωρών να προστατεύουν και να ενισχύουν τους εθνικούς τους πρωταθλητές εντός εισαγωγικών. Έτσι έρεται ένα εμπόδιο. Ολοκληρώνοντας μια τελευταία σκέψη, γνωρίζω ότι αυτές οι νησίδες συνεργασίας ίσως σας φανεί ότι είναι κατά της ιδέας μιας ε, πιο ενωμένης Ευρώπης. Όχι όμως, δεν πρόκειται γι' αυτό. Μιλώ για περιφερειακέ νησίδε συνεργασία, αναγνωρίζοντα τρει τρεις πραγματικότητε. Πρώτον, τα μεμονωμένα κράτη θέλουν να διαρθρώσουν τι στρατιωτικέ του δυνάμει όπω αυτά κρίνουν. Υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των διαφόρων περιοχών σε ό,τι αφορά τι ανάγκε και σε ό,τι αφορά τι δυνατότητε. Επίση, θα πρέπει να λυθούν υπόψη οι περιφερειακέ ιδιαιτερότητε αλλά και οι περιφερειακέ ομοιότητε. Άρα, νομίζω ότι η περιφερειακή προσέγγιση είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση για να έχουμε πρόσωπο τομέα του pooling και sharing και οι συμμετέχουσε χώρε έτσι θα γίνουν πιο ισχυρέ από στρατιωτική πλευρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόσβαση σε περισσότερε και όχι λιγότερε δυνατότητε στο μέλλον. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Μουρ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το όνομά μου είναι Graham Νιούρ, είμαι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και όπως τα άλλα μέλη του πάνελ δεν είμαι ακαδημαϊκός, δεν προέρχομαι από ένα think tank, είμαι εκπρόσωπος μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Ίσως επομένως να είμαι να, να μην είμαι πιο πρακτικός ε, από ότι οι άλλοι ομιλητές. Θα σας πω λίγα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε ε, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στο pooling and sharing. Γνωρίζετε ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ο διευθυντής μας, ο καινούριος διευθυντής μας πριν από μερικούς μήνες είχε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Το pooling και sharing, είναι, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας για την Ευρώπη. Και όπως είπε και ο στρατηγός Κούλμανς, δεν είναι κάτι το καινούριο. Εδώ και αρκετό καιρό το συζητάμε. Η υπηρεσία άμυνας δεν ευθύνεται εκείνη για το ότι η ιδέα αυτή υπάρχει εδώ και καιρό. Αλλά ε, από την δημιουργία της υπηρεσίας αυτής προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτή την ε, ιδέα της κοινή εκμετάλλευσης σε πολλούς τομείς και θα σας ε, ε, παρουσιάσω ποια είναι η κατάσταση για αυτήν την υπηρεσία μας που έχει 140 άτομα προσωπικό και όχι ιδιαίτερα μεγάλο προϋπολογισμό. Οι πρωτοβουλίες αυτές για το pooling και sharing δημιουργήθηκαν από ανάγκη και ήταν πρωτοβουλίες ad hoc κυρίως. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα να κάνουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι να δούμε αν μπορεί να γίνει μια πιο δομημένη προσέγγιση. Δεν αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι οι απόψεις των δύο προηγουμένων ομιλητών δεν αποκλίνουν μία την άλλη και νομίζω ότι θα μπορέσω να το αποδείξω. Ένα πράγμα είναι σαφές. Ούτως ή άλλως η άμυνα είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πάρουν την απόφαση για το κατά πόσον θα υπάρχει αυτή η συνεκμετάλλευση, ε, θα εφαρμόσουν δηλαδή την ιδέα του pooling και του sharing και με ποιον. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο θα το εφαρμόσουν όλοι. Και εδώ ε, θα μπορούσε να βοηθήσει βέβαια η υπηρεσία μας και θα σας εξηγήσω πώς πιστεύουμε εμείς ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. κατάρχα ο οργανισμό μας, η υπηρεσία μας, είναι μόνη, ο μόνος οργανισμός ο οποίο αναφέρεται στι ευρωπαϊκέ συνθήκε και ο μόνος και ε, ε, μόνη υπηρεσία όπου η Διευθυντική Επιτροπή συνεδριάζει σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Επομένως έχουμε θεσμικά μια μοναδική θέση και έχουμε και μεγάλη πολιτική προβολή. Επίσης ασχολούμεθα με όλο το φάσμα της δυνατότητας ε, ικανοτήτων, ε, δηλαδή κάνουμε μελέτες ε, και ανάπτυξη ικανοτήτων, βιομηχανική συνεργασία και θα ασχοληθώ με την βιομηχανική συνεργασία αργότερα. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, ο οργανισμός μας είναι ευέλικτος, δεν είναι ιδιαίτερα βαρημένη η η δομή του. Ε, ασχολούμεθα με δύο ειδών project. Το ένα είναι η δυνατότητα opt-out, δηλαδή ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν εκτός να αποφασίσουν να αποχωρήσουν και ένα άλλο μοντέλο είναι το opt-in, όπου απαιτεί, απαιτούνται δύο κράτη-μέλη για να ξεκινήσει η πρωτοβουλία και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη συμμετέχουν αν και εφόσον το επιθυμούν. Αυτό το οποίο εδώ αποδεικνύουμε είναι ότι έχουμε μία προσέγγιση à la carte, δηλαδή ε, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα ε, κάποιου κράτους μέλους, αποφασίζει το κράτος μέλος σε τι βαθμό θα συμμετέχει σε κάποιες βασικές μας εργασίες. Και αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει το pooling και sharing ε, ε, όπως είναι ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι καινούριο για μας, έτσι λειτουργούμε ούτως ή άλλως. Και είμαστε το ευρωπαϊκό κέντρο, αν θέλετε, του pooling και sharing. Έχουμε ξεκινήσει διάφορα project, ε, κάποια από τα οποία εξελίσσονται, προσφέρουν ε, βασικές ικανότητες σε μέρη όπου απαιτείται ε, να γίνει σοβαρή δουλειά, όπως προς χάρη στο Αφγανιστάν ή στα εργαστήρια που ε, εργαζόμαστε για τα, για τα εκρηκτικά. Είναι κάποια project αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή μας απασχολούν. Το πιο φιλόδοξο είναι ο, ο Ευρωπαϊκός Στόλος Αερομεταφορών. Ο δόκτωρας Βάλατσεκ αναφέρθηκε στην σημασία της βιομηχανίας και στην σημασία της συμμετοχής της βιομηχανίας. Εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό σαν βασικής ε, σημασίας θέμα. Δεν έχουμε μία απάντηση, αλλά ξέρουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχει η βιομηχανία και πριν από μερικούς μήνες ούτως ή άλλως οργανώσαμε ένα workshop με την βιομηχανία όπου εξετάσαμε τις συνέπειες που έχει το pooling και sharing στην βιομηχανία. Υπάρχουν θετικές συνέπειες βέβαια. Αν μια ομάδα κρατών μελών αποφασίσει συλλογικά ότι θα, χρησιμοποιήσουν από κοινού κάποιες υπηρεσίες υποστήριξης, τότε ο οργανισμός μας, οι υπηρεσίες μας μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη το catering, ε, μπορεί να φαίνεται ίσω μπανάλ το όλο θέμα, αλλά όπως είπε ο κύριος Βάλεσεκ, δεν ε, μιλάμε για ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία, αμυντική, στρατιωτική τέλο πάντων. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε ποιε είναι οι οικονομίες που θα μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι ώστε αυτοί οι περιορισμένοι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μα να χρησιμοποιούνται με, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μπορούν να ε, αναπτύσσονται οι δυνάμεις μας στα επικίνδυνα θέατρα του πολέμου. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή η κοινή χρησιμοποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με την συνεργασία. Ξέρω ότι αυτό είναι το βασικό θέμα, όχι του μήνα αλλά και ολόκληρου του χρόνου. Αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε σαν ζωτική σημασία είναι ότι όσο περισσότερο εφαρμόζεις αυτή την, ε, την ιδέα του pull share, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είσαι. Και αυτό είναι σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη μας ε, τα, το διαφορετικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη στις διάφορες επιχειρήσεις που δεν είναι διαλειτουργικό αν θέλετε. Και πιστεύουμε ότι αν υπάρχει αυτή η ιδέα της κοινή χρησιμοποίησης, η κοινή εκμετάλλευσης, τότε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας γιατί είναι πρώτη γραμμή αν θέλετε. Τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα για την υπηρεσία μας οι Υπουργοί ε, συναντήθηκαν στις 23 Μαΐου στην, στα πλαίσια της Διευθυντικής Επιτροπής και μας ζήτησαν να κάνουμε αυτό το οποίο ζήτησε ο καθηγητής κ. Βάλοτσεκ. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και να διδαχθούμε από τα παθήματα αλλά και από τις επιτυχίες των προηγουμένων εμπειριών που αφορούν αυτή την κοινή χρησιμοποίηση, το pooling και sharing. Άρα με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προσφέρουμε, να υποβάλουμε στα κράτη-μέλη προτάσεις ε, για το τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι είναι απόλυτη καταστροφή. Αν και απόλυτες καταστροφές λίγες έχουμε να κάνω δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις ε, υπομορφή συμπερασμάτων τελειώνοντας. Όπως ανέφερα πριν από ένα λεπτό περίπου, η υπηρεσία μας ε, πιστεύει ότι μπορεί να άρει κάποια από τα εμπόδια που αφορούν την κοινή χρησιμοποίηση, κοινή εκμετάλλευση ε, εντοπίζοντας τα παθήματά μας του, παρελθόν, του διότι δεν έχουμε εντοπίσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, όλες τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάποια εγκάρσια προβλήματα, π.χ. την ασφάλεια των προμηθεών. Αυτό όμως το οποίο είναι σαφές είναι ότι για να μπορέσουν να, να, μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά, και αυτό είναι κάτι το οποίο είπε και ο στρατηγός Κούμων, είναι ότι ε, χρειάζεται πολιτική στήριξη και πολιτική προώθηση η οποία θα είναι σταθερή και στο υψηλότερο επίπεδο. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάφορα θέματα. Ε, δεν, θα, δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα πάντα. Ε, η υπηρεσία ανήκει στα κράτη-μέλη. Ο προϋπολογισμός μας προέρχεται κατά 100% από τα 26 συμμετέχοντα κράτη-μέλη δεν είμαστε ένα υπεραθνικό σώμα, έχουμε μετόχους αν θέλετε. Και αυτό το οποίο ε, θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Αλλά τελικά οι επιλογές για το pooling και sharing, για αυτή την κοινή εκμετάλλευση, κοινή χρησιμοποίηση, είναι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν τα κυρίαρχα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις σε σχέση με τις... Εσείς παρακαλώ, έχετε τον λόγο, ζητώ συγγνώμη. Uh, ναι, καταρχήν ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ τους τρεις εισηγητές. Σημείωσα αρκετά πράγματα. Αυτή την ακρόαση την έχουμε υπόψη ως μια, ένα πρώτο βήμα για την εκπόνηση μιας έκθεσης στην υποεπιτροπή μας. Έτσι λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία για προβληματισμό. Food for thought έχουμε εδώ σε σχέση με τις, ε, τα διαφορετικά, τις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τα όρια που υπάρχουν όπως παρουσιάστηκαν. Και έχουμε και τις βέλτιστες εναλλακτικές προοπτικές ή δυνατότητες για αυτά τα οποία λειτουργούν, μπορούν να λειτουργήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα όλοι οι εισηγητές κατά κάποιο τρόπο ας το πω έτσι σκιαγράφησαν τις προοπτικές ίσως των παλαιών κρατών μελών και ξέθεσαν αυτές τις προοπτικές. Και είναι ενδιαφέρον ότι καμιά φορά νεότερα κράτη-μέλη είναι πιο φιλόδοξα από τα παλαιότερα κράτη-μέλη που έχουν παρακολουθήσει αυτά τα πράγματα επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε ότι νέα, νεότερα κράτη-μέλη είναι πιο φιλόδοξα και μπορείτε, μπορείτε υπό το πρίσμα το αυτό για την Πολωνική Προεδρία να, ελπίζει, να ελπίζουμε κάποιες νέες πρωτοβουλίες. Από τη μία ή άλλη πλευρά, από, τις Πολωνική, από την Πολωνική πλευρά κάποιες παρεμβάσεις ε, γίνονται ή μπορούν να γίνουν ώστε να υπάρξει ένα πιο φιλόδοξο επίπεδο στο επίπεδο του Συμβουλίου με την Πολωνική Προεδρία. Τις συμπράξεις και τις κοινέ αυτές δράσεις pooling and sharing τις αναφέρατε σε ένα κοινό επίπεδο για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Στην πρακτική εφαρμογή είναι όμως ε, διαφοροποιημένα τα πράγματα, διαφοροποιούνται. Πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό με την μία, με το pooling ή το sharing, με τις συμπράξεις ή τις κοινέ δράσεις, με τη μία ή την άλλη μπορεί να αναμένει κανείς περισσότερο ότι θα σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος σε σχέση για παράδειγμα με τις ε, συμπράξεις ή τις, ε, μια προσέγγιση όπου ένας έχει τα πάντα τα οποία διαθέτει και ο άλλος συμμετέχει επικερδός. Ε, και αποκομίζει κέρδος. Τι θα μπορούσε να είναι το πιο επιτυχές από αυτά τα παραδείγματα, ας το πούμε έτσι. Το πιο πολλά υποσχόμενο. Και εδώ ένα συγκεκριμένο ερώτημα που στο Ευρωκοινοβούλιο τίθεται για τα ευρωπαϊκά θεσμικά, για το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, το οποίο αυτό χρειάζεται συντονιστική δράση και που θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει προτάσεις για να προαχθούν τα πράγματα και όχι μόνο να συμπράττει απλώς παθητικά αλλά ενεργά Βλέπετε κάποιες περιφερειακές δυνατότητες ε, που μπορεί να δίνουν δυνατότητες. Απ' την άλλη πλευρά όμως ε, κάποιοι δεν θα θέλουν να περιοριστούν σε περιφερειακές δράσεις. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα. Υπό ευρωπαϊκό πρίσμα πρέπει να είμαστε πιο σφαιρικοί, πιο ολοκληρωμένοι και θα ελπίζαμε μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας ε, που πολιτικά η κυρία Άστον αναλαμβάνοντας δράσεις με συγκεκριμένες προτάσεις που θα είχαμε για την περαιτέρω πορεία μας. Δεν θα τα αφήναμε τα πράγματα στην τύχη ή στην συγκυρία για τα όσα θα γινόντουσαν από τα κράτη-μέλη. Βλέπετε εκεί τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας υπό τον όρο να υπάρχει πολιτική βούληση, κυρίως από την κυρία Άστον. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο παρακαλώ εσείς να απαντήσετε. Κυρία Κόμες, για το ερώτημα αυτό το οποίο μόλις έθεσε ο κύριος Γκάλερ και εγώ θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι στις ε, αμυντικές αγορές αμυντικού υλικού αυτό έχει κέρια σημασία όχι μόνο για τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Βάλασεκ ε, για τα όσα συμβαίνουν στον τομέα των κοινών δράσεων και συμπράξεων. Αλλά έχουμε αυτή την οικονομική κρίση με τεράστια ελλείμματα πολιτικά και οικονομικά για τη δράση μας, για τη χρηματοδότηση των ε, αμυντικών δράσεων και της, ε, στον τομέα ασφάλειας. Και ως πολιτικοί δεν μπορούμε να στραφούμε στους πολίτες μας και να απαιτήσουμε να χρηματοδοτήσουν την άμυνα και την ασφάλεια αν ε, θα θεωρούν ότι αυτό δεν είναι το πιο αποτελεσματικό. Και όταν υπάρχει τέτοια διαφθορά στη χώρα τη δική μου, στην Πορτογαλία, όλες οι δημόσιες προμήθειες βρισκόντουσαν υπό την απειλή της διάβρος, της ε, διαφθοράς και δεν είναι πορτογαλικό, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Βλέπουμε και σε σχέση με τη Γερμανία ή τη Γαλλία ή τους Αμερικανούς είναι πραγματικό πρόβλημα το θέμα της διαφθοράς. Αυτό είναι κέρια σημασία ζήτημα και πρέπει σε σχέση με τους πολίτες μας να το αναγνωρίσουμε όταν ζητάμε να υποστηρίξουν τέτοιες δράσεις και ζητάμε <clears throat> από πλευράς των πολιτών να διατεθούν κονδύλια για τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ασφάλειας. Θα ήθελα λοιπόν τούτων λεχθέντων να σας ρωτήσω κάτι. Από όλους αυτούς τους τομείς και τα πεδία αυτά που εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν ως προτεραιότητες για τις κοινέ δράσεις και τις συμπράξεις ε, για τον τομέα άμυνας. Ποιοι είναι εκείνοι οι τομεί όπου υπήρξε κινητοποίηση, ποιοι είναι εκείνοι οι τομεί και τα πεδία όπου τίποτα δεν έγινε και ποιοι θα έπρεπε να είναι πραγματικά η προτεραιότητα στην οποία θα επικεντρωθούμε σε αυτή τη φάση. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φυσικά γνωρίζω, γνωρίζω ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία αναγνωρίζω τις ανησυχίες για να υπογραμμιστούν αυτά τα θέματα, ότι τίποτα δηλαδή δεν θα γίνει κατά της εθνικής, των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν θα ήταν όμως λογικό να ζητούσαμε από τα δύο κράτη-μέλη εκείνα τα οποία διαθέτουν περισσότερα στην άμυνα και την ασφάλεια μικροφωνισμός από πλευράς της ομιλήτριας ή του τηλεφώνου της δεν θα έπρεπε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει έναντι άλλων που δεν ε, δρούν παράλληλα. Θα λέγατε ότι η τελευταία αυτή γαλλοβρετανική συμφωνία για τα θέματα άμυνας αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλα τα κονδύλια που διατίθενται στον ε, πυρηνικό τομέα ε, ουσιαστικά δεν έχουν αντίκρισμα. Και σε σχέση με τον κύριο Μόερ εν τέλει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, να μην έχουμε κονδύλια για την ε, επάρκεια που απαιτείται λόγω της οικονομικής κρίσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Ποιες είναι οι προοπτικές έναντι για παράδειγμα των Κινέζων που εξαγοράζουν ευρωπαϊκές εταιρείες και το χάσμα τεχνολογίας ε, που υπάρχει και δημιουργείται σε σχέση με την Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Um, thank you, Mr. Κάμπλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το πάνελ ε, γιατί ήταν πάρα πολύ ε, μεγάλη εμπειρία που έδειξαν ε, με τις ομιλίες του σήμερα, καταφέραμε να μην αναφέρουμε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό οργανισμό που έχει τα όμως ε, την έδρα εδώ στη Βρυξέλλες και που είναι πολύ καλός στο σε το ΝΑΤΟ δηλαδή. Θα ήθελα να ξέρω τις απόψεις των μέλων του πάνελ. Αν δεν υπάρχει πολύ χρήμα, το είπαμε αυτό, και αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε πόρους, μήπως θα έπρεπε να αποφεύγουμε αυτή την επικάλυψη σε αυτές τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και πράγματι υπάρχει αυτή η αλληλοεπικάλυψη σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα με ενδιαφέρει να μάθω αν θεωρείτε ότι κάποιε από τι πρωτοβουλίε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλληλοεπικαλύπτουν και μάλιστα υπονομεύουν ε, τι επιχειρήσει του ΝΑΤΟ και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα του κόστου και πώ θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Τα μέλη του πάλι για να απαντήσουν. Κύριος Κόλμαντ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω αντί, ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Μιλήσαμε για το pooling και sharing και νομίζω ότι και εγώ αναφέρθηκα στην ομιλία μου στο γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΝΑΤΟ και κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Είπατε επίσης ότι ο είναι πολύ καλό στο pooling και sharing. και καλό θα ήταν να το ακολουθήσουμε κι εμείς και αυτό καλό θα ήταν. Ξέρουμε ότι δεν είναι υπερεθνική οντότητα ο οργανισμός αυτός και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο πιο μεικτή, άρα αν γίνει κάτι στο ΝΑΤΟ γίνεται γιατί θέλουν να γίνει οι χώρες μέλη του. Και πράγματι υπάρχει καλό pooling και sharing, υπάρχουν και τα θέματα της τυποποίησης που έχουν πολύ καλές εξελίξεις και πολύ καλές ε, είναι και επαφές των δύο οργανισμών. οι Ρέψ, η στρατιωτική ε, αντιπρόσωπη του ΝΑΤΟ είναι και στρατιωτική αντιπρόσωπη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λήφθη μια απόφαση ότι τα πρότυπα που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ είναι τα ίδια τα οποία χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων. η μόνιμη έδρα, το μόνο στρατηγείο επίσης είναι κάτι πολύ καλό και είναι λογικό. Αν κάποιο θέλει να κάνει στρατηγική επιχείρηση, το πρώτο στοιχείο είναι να είναι μόνιμη στρατηγική έδρα, όπως γίνεται με τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ επίσης, που έλαβαν τη σοφή απόφαση να έχουν ένα επιχειρησιακό στρατηγείο. Ενώ εμείς έχουμε 5-6 και κανένα μάλιστα δεν ε, λειτουργεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε ένα μόνιμο επιχειρησιακό στρατηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλό επίσης είναι να, έχουμε, ε, να συνεχίσουμε να έχουμε τον καλό διάλογο με ταξί Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε ερωτικό επίπεδο. Ξεχάστε αυτό ότι το παλιό απόθεμα ότι πρέπει να επιλέγουμε και ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ είτε ΝΑΤΟ είτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε για δυνατότητες. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Και βλέπουμε επίσης τα ελλείμματα, τις ελλείψεις που έχουμε όλοι, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δυνατοτήτων. Πραγματικά υπολοιπόμεθα στον τομέα αυτό και σε στρατηγικό επίπεδο. Πρέπει να υπερβούμε τις δυνατότητες της κάθε μιας μονομένης χώρας. Άρα όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε αλλιώς θα αποτύχουμε ε, χωριστά ο ένας ε, από τον άλλο. Επίσης πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική ξεκάθαρη και θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος οργανισμός ή πιο, πιο καλός φορές για να αντιμετωπίσει μια κρίση των αυτή προκύψει. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως κάνουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σε πλαίσιο κάποιων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, λοιπόν σε καμία περίπτωση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα δεν υπάρχει καν άλλη επικάλυψη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πολύ σοβαρή συνεργασία. Και ήδη το έχουμε πράξει και έρχομαι στο ερώτημα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Στο πλαίσιο τη σύμβαση σε, σε αυτό εδώ το κτίριο Τη συνέλευση που έγινε, ξέραμε πολύ καλά ποιε είναι οι δυναμίε μα. Και ξέραμε ότι χρειαζόμαστε κάτι σαν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Ο στόχο του δεν ήταν να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τακτική ή τα τεχνικά ζητήματα. Είχαμε απόψε μια πάρα πολύ καλή εξήγηση για τις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Λυπάμαι όμω, αλλά είχαμε λαμπρά παραδείγματα σε επίπεδο τακτικής, ε, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να έρθουμε στο ε, επίπεδο των προσδοκιών μας. Δεν φταίει ο οργανισμός άμυνας βέβαια. Το θέμα είναι ποιος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είπατε εκπρόσωπος είναι ε, η Προεδρεύουσα και οι υπόλοιποι είναι Υπουργοί Άμυνας. Άρα αυτοί είναι που έχουν την αρμοδιότητα. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση της κατάστασης. Γιατί υπάρχει ομοφωνία αυτή τη στιγμή. Αν αρνηθεί μια χώρα δεν γίνεται τίποτα και δεν σημειώνεται πρόοδο. Ίσως υπάρχουν χώρε που θέλουν να προχωρήσουν λίγο περισσότερο και λίγο πιο μακριά. Πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τέλο, και πάλι επαναλαμβάνω, σε εμά εδώ είναι απόκτηση στην Ευρώπη. Ας ε, ανταποκριθούμε στι προσδοκίε μας, στις φιλοδοξίες μα και α χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία έχουμε ήδη αναπτύξει για το στόχο που τα έχουμε αναπτύξει. Τελευταίο στοιχείο ο Γκάλερ το ανέφερε, πούλινγκ και sharing. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε και την εξειδίκευση, το specialization. Και όλα αυτά είναι ένα τρίο, μια τριάδα που παράγει όφελος. Πρέπει να καταλάβουμε, ε, αν καταλάβουμε καλά το pooling, μπορούμε να κάνουμε και sharing. και μπορεί κανεί να μην είναι κοντά ε, γεωγραφικά με τον άλλο, μπορεί να έχει την ίδια προσέγγιση, την ίδια στρατηγική. Και φυσικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εθνική κυριαρχία με αυτή τη σύμπραξη, την κοινή εκμετάλλευση, γιατί είμαστε σε μια κοινότητα και μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξειδίκευση, χωρί κανένα πρόβλημα. Απλά πρέπει να φροντίσουμε να μην οδηγηθούμε στην κατεύθυνση τη εξειδίκευση αλλά με εθνική βάση. Γιατί τότε κάθε έθνο θα έχει το βέτο και αυτό θα δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε και την ειδίκευση σε αυτό το τρίγωνο. Διαφορετικά στοιχεία απαρτίζουν αυτό το τρίγωνο, υπάρχουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις για τη συνεργασία μεταξύ χωρών, αλλά όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους και νομίζω ότι τελικά αυτά τα τρία στοιχεία, pooling, sharing, specialization, είναι αυτά στα οποία αποσκοπούμε, αλλά ας αρχίσουμε με, όχι με τόσο μεγάλη βιασύνη. Αυτό το οποίο ε, υπόσχεται πολλά είναι η περιφερειακή διάσταση του pooling και sharing, αυτές είναι οι σύνδεσεις συνεργασίας. Ναι, ωραία. Αν αυτό το βήμα πρέπει να γίνει τώρα, ας γίνει. Και αν αυτό μας φέρει μπροστά, ας το κάνουμε. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι στρατηγικές μα ελλείψει. Και αυτό είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο πια στη διάθεσή μα. Όταν ήμασταν τότε, όταν επιχειρήσαμε στην πρώην Ιουκοσλαβία, πάλι το σκεφτόμαστε αυτό το θέμα των στρατηγικών ελλείψεων. Είχαμε μια δεκαετία μπροστά μα, τώρα όμω δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το μακροπρόθεσμο έγινε βράχη πρόθεσμο και είναι σήμερα. Next, please. Ο κύριος Βάλασεκ, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω εκεί που ο στρατηγός σταμάτησε. Το θέμα του δυναμικού σε σύμπραξη και κοινέ δράσεις περιφερειακά και με τις δυνατότητες αυτές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επί του θέματος αρχής αυτό που ζητείτε είναι η δημιουργική δυνατότητα εκμετάλλευσης, σύμπραξης και κοινών δράσεων. Και στη Λιβύη αυτό καταδεικνύεται. Να δούμε τη δυνατότητα που μπορούμε να δραχθούμε αυτή και να δράσουμε με μια κοινή, ε, σε μια κοινή βάση όλοι. Αναγνωρίζοντας ότι είναι φθηνότερο να το κάνουμε αυτό ε, σε σύμπραξη και κοινέ δράσεις από ότι ατομικά. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα δαπάνης νέων κονδυλίων σε αυτές τις δράσεις. Αυτή δεν είναι όμως η πραγματικότητα στην οποία ζούμε σήμερα. Η πραγματικότητα είναι περικοπές δαπανών για τα αμυντικά 50% για παράδειγμα, στον αφορά τη Λετωνία κάνουμε λόγο για σημαντικές περικοπές. Δεν υπάρχουν νέα κονδύλια λοιπόν να επενδυθούν. Γι' αυτό η περιφερειακή προσέγγιση ίσως είναι μία από τις καλύτερες δυνατότητες αναπτυξιακά να δούμε την προοπτική αυτή. Είναι απλή η προσέγγιση. Να δούμε τις ε, υποδομές ε, των δυνατοτήτων που έχουμε σήμερα και να τις χρησιμοποιήσουμε με πιο ευφυή τρόπο. Βλέποντας στην κεντρική Ευρώπη ότι δύο-τρεις χώρες ε, έχουν τις ίδιες κοινέ δράσεις, πρέπει μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο να δράσουμε. Και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ένα κέντρο μεταξύ αυτών των χωρών όπου θα επενδύαμε από κοινού. Να χρησιμοποιήσουμε το κοινό δυναμικό ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους, κονδύλια από τις υποδομές. Και όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες, νέο δυναμικό και θα δούμε και νέες ε, προοπτικές. Διαφορετικές χώρες θα θέλουν να αγοράσουν διαφορετικό ε, ε, εξοπλισμό. Δεν είναι όλα αυτά ασύμβατα. Πρέπει να δούμε σε κλιμακού προηγούμενη προοπτική την ανάπτυξή τους και για το, την δυνατότητα συνεισφοράς όσον αφορά το ε, ΝΑΤΟ έχω ε, μια ξεχωριστή προσέγγιση που θα ε, υποβάλω και στους επικεφαλείς του ΝΑΤΟ. Αλλά υπό αυτό το πρίσμα κάθε θεσμικό όργανο έχει συμπληρωματική δράση έναντι του άλλου και μπορεί έτσι συμπληρωματικά ή παραπληρωματικά να δράσει. Και σε σχέση με την ε, ε, παρέμβαση σε σχέση με το ΝΑΤΟ και το δυναμικό του με την ε, εκπόνηση των ερωτηματολογίων ή την ε, δυνατότητα ανείχνευσης των δυνατοτήτων μπορούμε να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν περιφερειακά. Το ΝΑΤΟ κινήθηκε και στην περιφερειακή διάσταση. Αντί να λέμε σε επιμέρους χώρες το τι μπορούν να αγοράσουν, περιφερειακά θα είναι δυνατόν να δράσουμε. Είναι μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα να κινητοποιηθούμε ώστε να μπορέσουν οι χώρες να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης μέσα ε, ε, για παράδειγμα της προσπάθειας κοινή χρήσης ε, κοινών δυνατοτήτων σε σύμπραξη και κοινέ δράσεις. Μπορούμε έτσι μέσα στο πλαίσιο αυτό να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από πλευρά των δράσεών μας. Η θετική επικάλυψη, ας την αποκαλέσουμε έτσι, positive duplication, η έχει θετικές επιπτώσεις. Τώρα για το θέμα της διαφθοράς θα πρέπει να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις της κυρίας Γκόμε. και βλέπουμε ότι σε σχέση με τη διαφθορά το ε, ποσοστό σε σχέση με τις ε, ε, του 2% ε, αν το ποσοστοποιήσουμε σε αυτό είναι πραγματικά ε, μειώνει τις δυνατότητές μας. Θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε ποιοτικά και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε ε, με ιδιαίτερη προσοχή. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι κάτι το οποίο το αφήνω σε εσά και να δούμε το ρόλο του ΝΑΤΟ, το, την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ε, ΝΑΤΟ δυνατότητες ε, σε κοινή δράση μεταξύ, των, ε, μεταξύ κάποιων χωρών. Είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε και να μας απασχολήσει. Μια τελευταία παρατήρηση για ένα τελευταίο θέμα και ζητώ συγγνώμη αν δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις αν το pooling και sharing θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη των νεότερων κρατών μελών και με ένα πιο φιλόδοξο τρόπο. Οι ιστορίες των επιμέρους κρατών μελών είναι ε, ε, διαφοροποιούνται μεταξύ τους και πρέπει να δούμε το πώς οι ομάδες, οι μάχημες ομάδες θα μπορέσουν να προσαρμοστούν είναι ένα από τα πιο συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να προσφέρει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στις νεότερες χώρες για αυτές τις δράσεις με ε, τις επαφές με τους ε, συναδέφους ε, σε σχέση με την ε, Πολωνία, με την αξιολόγηση των κοινών δράσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την, τον κοινό προβληματισμό και την δραστηριοποίηση βλέπουμε τις χώρες Μπενελούξ, τις σκανδιναβικές χώρες, την πρόσφατη περίπτωση της γαλλοβρετανικής συνεργασίας που και σήμερα ακόμα μπορεί να ε, προσφέρει δυνατότητες ε, το pooling και sharing. Βλέπουμε οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι ε, εξετάζουν και διερευνούν αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχει δυναμικό. Η κυρία Γκόμες θα είναι σε καλύτερη θέση να μας αναφέρει τα, σε σχέση με την Πορτογαλία αλλά φυσικά υπάρχουν περιθώρια για να μπορέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα των κοινών δράσεων και συμπράξεων να προαχθεί. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πάσκου, παρακαλώ. Um, Θα ήθελα να συγχαρώ το πάνελ για τον επαγγελματικό τις επαγγελματικές τους ικανότητες και τις ομιλίες οι οποίες προκάλεσαν ε, όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δεν συζητήσαμε πολύ παραπάνω από το pooling και sharing. Και αυτό το pooling και sharing ε, παρουσιάζεται μέσα από το παράδειγμα συνεργασίας Γαλλίας και Ενωμένου Βασιλείου, που είναι μια ειδική περίπτωση, δεν μπορεί να γενικευθεί εύκολα. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι λογικό. Ξέρετε ότι η περιφερειακή προσέγγιση είναι λογική, είναι σωστή. Η ανάγκη να έχουμε παρόμοιες κουλτούρες είναι κάτι σωστό. Ε, εδώ και χρόνια, εκατοντάδες χρόνια η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο είχε κάποια συνεργασία ε, ενώ είχε πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία με τη Γερμανία ε, που ήταν η πυρωτική χώρα. Το Βέλγιο και η Ρουμανία έχει επίσης κοινά στοιχεία, ε, βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Ίσως το Βέλγιο είναι λίγο πιο πάνω από μάσα. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει μια ήπειρος που μας χωρίζει. Είναι τελείως διαφορετικές οι παραδόσεις. Επομένως επανερχόμεθα στο θέμα των διαφορών ανάλογα με τις περιοχές. Όμως, τι συμβαίνει. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι και ασχολούμεθα με τα εσωτερικά μας θέματα και εσωτερικές μας υποθέσεις και αγνοήσαμε το, το γεγονός ότι έπρεπε να διατηρήσουμε τις επαφές μας με άλλες χώρες, με την, στην περιοχή μας ενδεχόμενα έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό παρονομαστή όσον αφορά την αντιμετώπιση κάποιων ε, καταστάσεων. Ξέρω ότι η Γαλλία και το Αναμένο Βασίλειο αντιμετώπισαν τα προβλήματα στην Λιβύη. Κάνανε αυτή την κοινή χρησιμοποίηση, κοινή εκμετάλλευση ε, για ε, να οργανώσουν αυτή την κοινή επιχείρηση κατά των δυνάμεων του Καντάφη. Στη δική μας όμως περιοχή η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και άλλες χώρες, ας πούμε στα Δυτικά Βαλκάνια, η πιο στο βορρά η Ουγγαρία, τι πρέπει να κάνουνε. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό πιστεύω. Θα πρέπει να επανεστιάσουμε την προσοχή των ηγετών των χωρών στην ανάγκη που υπάρχει να επενδύουμε στην άμυνα. Πρέπει να προσέχουμε την άμυνα. Έχουμε στοιχεία ε, στο παράρτημα εδώ που σταματούν στις αρχές του 2010. Έκτοτε η κατάσταση βελτιώθηκε, επιδεινώθηκε θα έλεγα. Μία χώρα η οποία ενθαρρύνει τις μειονότητες που ζουν σε άλλες χώρες γειτονικές να αντιμετωπίσουν ε, ε, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τη χώρα στην οποία να ζουν. Αυτή η χώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα. Τέλος πάντων θα πρέπει να σκεφτούμε συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο έτσι ώστε και οι κάτοικοι και ο πληθυσμός να το συνειδητοποιήσει γιατί και ο πληθυσμός και οι πολίτες θα ε, ταρακουνήσουν τους ηγέτες, τους πολιτικούς ηγέτες έτσι ώστε να προσέξουμε την άμυνα. Όταν συζητάμε για τις περιφέρειες θα πρέπει σοβαρά να λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιφερειών ε, όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε είναι φυκτά και αν ναι διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν χάσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν τα κράτη-μέλη τους έτσι ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν όλοι στην διατήρηση ενός συγκεκριμένου επίπεδου της ασφάλειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μούρ Ευχαριστώ. Τέσσερις, τέσσερα ερωτήματα νομίζω τέθηκαν άμεσα προσωπικά σε μένα. Αν αμελήσω κάποιο, οπωσδήποτε θα μου το υπενθυμίσετε σίγουρα. Ξεκινώντας με το ερώτημα για τον ΝΑΤΟ, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτή την παρατήρηση και σίγουρα πράγματι θα πρέπει να το είχα αναφέρει, αλλά το αμέλησα. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την παράληψη. Όμως εμείς ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα συνεργαζόμαστε στενά με τον ΝΑΤΟ. Ακριβώς επειδή πρέπει να διασφαλίζουμε ότι το έργο μας θα είναι παραπληρωματικό, συμπληρωματικό και σε σχέση με ε, τις προσπάθειες που ε, καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε σχέση με το δυναμικό θα πρέπει και σε σχέση με συ, συμμαχικές δράσεις να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ιδιαίτερα για την ε, δεν χρειάζεται να ε, πηγαίνουμε στο Norfolk της Virginia. Υπάρχει γραφείο στο Shape, στο Mons, στο Βέλγιο και βρισκόμαστε σε άμεση επαφή. Το σημαντικό θέμα που πρέπει να τονίσουμε δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να αποφεύγουμε διπλοεπικαλύψεις, αλλά να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν κενά, δεν θα υπάρχουν χάσματα. Και επειδή έχουμε κοινή ιδιότητα ε, που μας χαρακτηρίζει ως μέλη, τα περισσότερα ε, στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτά τα, αυτές τις δράσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο ΝΑΤΟ είναι ταυτόσημα. Και Πράγματα τα οποία ε, υπογραμμίζονται εδώ σε σχέση με τις δύο αυτές, ε, τα δύο θεσμικά αυτά όργανα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν είναι ένας διαγωνισμός, ε, ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει περιθώριο και για τις δύο οργανώσεις και για τους δύο οργανισμούς να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ατομικά και συλλογικά αποτελεσματικά. Δεν είναι λοιπόν σε ανταγωνισμό του ενός εναντί του άλλου και θα πρέπει αυτά όλα να αναπτύσσονται με ένα, σε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο. Για το επόμενο ερώτημα, κυρία Γκόμεσε, δεν είμαι βέβαιος ότι εγώ είμαι το πιο κατάλληλο άτομο να απαντήσω αυτό το ερώτημα όσον αφορά τις αγορές των Κινέζων στην Ευρώπη τεχνολογίας και βιομηχανιών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχουμε ε, υπαλλήλους Κινέζους ε, στο δικό μας ε, οργανισμό η βιομηχανική αυτή κύκλη είναι οι βιομηχανίες, οι αμυντικές βιομηχανίες και είναι αρμοδιότητα των εταιριών αυτών που ασχολούνται με την παραγωγή αυτού του υλικού. Δεν έχουμε υπόψη να έχουν αγοράσει οι Κινέζοι τέτοιες εταιρείες ή τέτοια τεχνολογία σε αυτό το ε, τομέα. Αλλά το κύριο ερώτημα είναι για τις προτεραιότητές μας. Δεν εργαζόμαστε σε στεγανό πλαίσιο, εν κενό ε, είναι ένα δυναμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσουμε τις ε, ε, προοπτικές και τις πρωτοβουλίες για το δυναμικό μας ε, και την ανάπτυξη του δυναμικού όπως το ανέφερε ο στρατηγός Κόλμαν πιο πριν. Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη σειρά προτεραιοτήτων μέσα στην προοπτική ανάπτυξη του δυναμικού μας και για αυτές τις προτεραιότητες καταβάλουμε προσπάθειες. Θα έλεγα όμως ότι δεν είναι το μόνο δόγμα αυτό, δεν είναι το κάτι το οποίο είναι θέσφατο και απαιτεί Τίτε η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των κρατών μελών και των συμφερόντων τους. Αλλά μέσα από πολλές πρωτοβουλίες ε, σύμπραξης και κοινών δράσεων από πλευρά ε, του οργανισμού μας ε, αναπτύσσονται στον άξονα του προγράμματος ανάπτυξης δυναμικού. Για παράδειγμα, οι δυνατότητες εναέριων μεταφορών και του στόλου εναέριων μεταφορών για την αποτελεσματικότητα της κάλυψης των αναγκών μας. Έχουμε ένα πλαίσιο δράσης ακόμα και όσον αφορά και τις επικοινωνίες με δορυφόρους. Και ακόμα και ένα άλλο ερώτημα νομίζω υπήρχε από τον κύριο Γκάλερ που τέθηκε για τον ρόλο της Κάθριν Άστον ως είπα της εκπροσώπου. Όπως θα γνωρίζετε η ε, Κάθριν Άστον έχει τρεις ιδιότητες. Η τρίτη της ιδιότητα πέρα από το ότι το τρίτο της αξίωμα, πέρα από το ότι είναι, είπατε εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι είναι επικεφαλής αυτού του οργανισμού και Ω επικεφαλής αυτού του οργανισμού και όπως ανέφερε και ο στρατηγός Κόλμοντ είναι επικεφαλής του Συμβουλίου μας για τα θέματα τα αμυντικά και ε, των αμυντικών πρωτοβουλειών αναφέρεται και υποβάλλει εισηγήσει στου υπουργού, υποβάλλει συστάσει πώ θα έπρεπε να αναπτυχθεί το έργο στο μέλλον. Φυσικά αυτό προϋποθέτει και ένα πλαίσιο συνένεση και συμφωνία. Διαδραματίζει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ρόλο η κυρία Άστον και το γεγονό ότι έχει αυτά τα τρία αξιώματα ή τι τρει ιδιότητε και υπό το δικό μου πρίσμα προσωπικά το αναφέρω αυτό, θεωρώ ότι είναι ζωτικού χαρακτήρα, έχει ζωτικό χαρακτήρα και είναι υποφελέ για μα, διότι εμείς στον οργανισμό μας δεν είμαστε μια απομονωμένη νησίδα. και όπως σε σχέση με τον κύριο ε, βάλασε και την παρέμβασή του, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αρκετούς τομείς και θέματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέργεια πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Άστον διευκολύνει αυτόν τον διάλογο που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί ενός ολοκλήρου φάσματος θεμάτων. για παράδειγμα, όσον αφορά τη συμφόρηση των ευρωπαϊκών ουρανών και των, ε, του συνοστισμού που σημειώνεται μέχρι και τις ε, δορυφορικές επικοινωνίες με αποτελεσματικό τρόπο επιλαμβάνεται των καθηκόντων της και μεριμνά ώστε οι υπουργοί να μπορούν να βρίσκονται στο αναγκαίο ε, επίπεδο και ενημέρωσης και συμμετοχής και παρέχει, παρέχεται έτσι και διασφαλίζεται η πολιτική υποστήριξη για αυτό το έργο που διασφαλίζει. Ευχαριστώ. Λίγα τελευταίες παρατηρήσεις από τον Δρ Μέλιγκερ και από τον Δρ Μάλι. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα σχόλια. Μου έρχεται να μπω στον πειρασμό να απαντήσω στην κυρία Γκόμες για τα περί διαφθοράς και για την ε, υπόδειξη να ρωτήσουμε τον κόσμο. Ίσως να είμαι κοινικός γιατί έχω εργαστεί πολύ για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αν ζητήσει κανείς ε, τους ντόπιου, ε, στα ναυπηγεία παραδείγματο χάρη, σε όποια χώρα θέλετε, και αν τους ρωτήσουμε αν νομίζουν ότι είναι καλό να ναυπηγείτε το ένα ή το άλλο πλοίο στα ναυπηγεία τους και αν η ε, πολιτική για αυτούς είναι καλή ή κακή, νομίζω ότι η απάντησή τους θα είναι δεν με νοιάζει ε, πώς θα έρθει η... ποια θα είναι η κατάληξη με ένα διαγωνισμό, ε, σε σχέση με τη δουλειά μου. Υπάρχει νομίζω κάποια συμμαχία. Ε, το θέμα είναι να πάρουν τη δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι διαφθορά. Ε, σίγουρα υπάρχουν και κάποια συμφέροντα που σχετίζονται και με την ασφάλεια. Τέλος πάντων υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Πάντως, γενικά συμφωνώ ότι είναι ένα πρόβλημα η διαφθορά με τις συμβάσεις, με τους διαγωνισμούς Αλλά τώρα κατά πόσο να ρωτήσουμε τον κόσμο για το τι ε, άποψη έγινε δεν ξέρω. Τώρα, σε ό,τι τον κύριο Γκάλερ, τη διαφορά στα επίπεδα φιλοδοξίας μεταξύ νέων και παλιών κρατών μελών, αν είναι πιο ενεργά η δραστήρια ή όχι, κάποιες φορές είναι. Αν δει κανείς στη Σουηδία, για παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση από διαρθρωτικής πλευράς με την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από στρατιωτικής πλευράς δεν έχει κάποια, κατανάγκη κάποιο νόημα, κάποια σημασία. Αν η δραστηριότητα είναι ο ρυθμός των συνασπισμών ή των δραστηριοτήτων που και θα δούμε ότι ένα από τους πιο δραστηριούς εταίρους είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι και πάρα πολύ προσεκτικό κράτο μέλο, αλλά και πολύ δραστήριο στον τομέα του pooling και sharing. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανεί έτσι πολύ ε, απλά με βάση δύο-τρει κανόνε και να αξιολογήσει και να υπολογίσει πώ λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Πολωνία φαίνεται να ε, γίνεται ένα ε, ηγέτη πλέον μεταξύ των πιο μικρών κρατών μελών και αναλαμβάνει τα ενία αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Θα ήθελα να διαφωνήσω με κάτι που φαίνεται να είναι πίσω από όλη τη σημερινή ε, συνάντηση, ότι η τακτική pooling και sharing οδηγεί σε οικονομίες. Δεν συμφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα το pooling και sharing, και αυτό πάντοτε προσπαθώ να το θυμίζω ε, σε ό,τι αφορά το κόστος μεταποίησης. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να υπάρχουν χρήματα, να υπάρχουν επενδύσεις. Με τις αμυντικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη, το περίεργο είναι ότι νομίζουν ότι μπορούν να μετασχηματίσουν ε, τον αμυντικό τους μηχανισμό χωρίς να κάνουν τίποτα. Μα πρέπει να έχεις χρήματα για να τα πετύχεις αυτά. Άρα, για να είναι βιώσιμο, ε, βιώσιμες οι κοινές δράσεις, και η συνένωση πόρων, όπως είπαν και προλαλήσαντες, χρειάζεται κανείς τη βιομηχανία, γιατί οι λύσεις είναι μακροχρόνιες λύσεις. Δεν μιλάμε για τον τάδε το δίνα εξοπλισμό και να κάνουμε πουλν και sharing σήμερα, αλλά μιλάμε για την μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης, κοινή ανάπτυξης πραγμάτων για να εξοικονομηθούν χρήματα. Η διαλειτουργικότητα είναι κάτι που συνεπάγεται πολλές δαπάνες. Πολλές εταιρείε προσπαθούν να αναπτύξουν πράγματα που να καθιστούν ε, μηχανήματα ή μηχανές ασύμβατες μεταξύ τους, να τι καταστούν συμβατές, να τι καθιστούν συμβατές. Ο κύριος Κάμπελ πάρα πολύ καλά τα είπε. Το ΝΑΤΟ είναι ένα σημαντικός παίκτη στον τομέα των δυνατοτήτων και τη ανάπτυξη δυνατοτήτων. Θα έλεγα όμως, υπάρχει και ένα φυσικό όριο στην δυνατότητα του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίζει τι σημερινέ προκλήσεις για τον απλό λόγο ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει μια βιομηχανική πολιτική, δεν έχει μια τεχνολογική πολιτική. Εμείς όμως, τουλάχιστον στην μη στρατιωτική διάσταση, το έχουμε αυτό. Και μέσω της Κομισιόν λοιπά Ίσως αυτό περάσει και στην στρατιωτική διάσταση. Αν ε, σκεφτούμε ε, με την ε, νοοτροπία των ΣΥΛΟ και αν σκεφτούμε τι θα μπορούσε η ανάπτυξη από, πλευρής, ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ωφελήσει το ΝΑΤΟ παραδείγματος χάρη. Αυτό ίσως θα έπρεπε να το δούμε. Κύριε Γκάλερ, το ερώτημά σας ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και κάποιες φορές χάνουμε την ουσία. Διότι έχουμε την, έχουμε την προσφορά και τη ζήτηση. Βέβαια δεν μου αρέσει ο όρος ε, μικρές ή μεγάλες χώρες, ε, αλλά πράγματι οι χώρες που δεν έχουν πολλά χρήματα να δαπανίσουν ενδιαφέρονται περισσότερο για την καινοτομία. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε μείωση των δαπανών αφενός αλλά αφετέρου έχουμε άτομα τα οποία προσπαθούν με λιγότερα χρήματα να βρουν λύσεις, όπως ε, είπε και ο προλαλής σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν πρέπει να είμαστε κοντόθωροι. Δεν μπορούμε να προασπίζουμε τα κεκτημένα και τα συμφέροντά μας. Υπάρχουν κάποιες μικρές χώρες που δεν έχουν δυνατότητες. Άρα τι πρέπει να κάνουν, δεν έχουν την παράδοση, δεν έχουν την κληρονομιά, μπορούν να καινοτομήσουν. Η Σουηδία, για παράδειγμα, μπορεί να καινοτομεί, μπορεί να είναι δημιουργική. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό. Και το χειρότερο θα ήταν να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της τόχιας της ε, διαχείρισης προσπαθώντας να μειώσουμε μόνο τις δαπάνες και διατηρώντας όλες τις δυνατότητες. Πρέπει να έχουμε μια, ένα πολιτικό όραμα. Να πιέσουμε προς μεγαλύτερη καινοτομία. Αυτό να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ένα στρατιωτικό οργανισμό ή να προσπαθήσουμε με μια αλωνιστική μηχανή να σταματήσουμε ένα τάγκ. δεν υπάρχει κατά ανάγκη αντίληψη της κατάστασης. Πρέπει να έχουμε όραμα. Το γαλλικό παράδειγμα είναι σημαντικό. Δεκαετία του 50. Συντηρητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τι αρχιωτικέ δαπάνε. Και εξάρτηση από τις ΗΠΑ σε σχέση με τη βιομηχανία. Και η βιομηχανία και η στρατιωτική αν τους ρωτούσε κανείς, ήθελαν να μείνουν εκεί τα πράγματα. αλλά είχαμε τον στρατηγό Ντεγκόλ που ε, δρομολόγησε κάτι καινούριο και οδήγησε όλους σε μια νέα συνένεση. Και ίσως κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρούμε ένα νέο όραμα. Θέλω να πω προς την κυρία Γκόμες ότι οι αποστολές είναι Πρόκληση είναι και ευκαιρία. Γιατί υπάρχει το κοινό όραμα. Σε ό,τι αφορά ε, τη γαλλογερμανική συνεργασία, αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να υπάρξει ένα κοινό όραμα. Να υπάρχει και η, επιθετική, η αμυντική και η επιθετική, αν θέλετε, προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη προσφορά Υπάρχει μονοπωλιακή κατάσταση της βιομηχανίας. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα διμερές μονοπόλιο όμως. Θα πρέπει να το διευρύνουμε όμως ε, το επίπεδο αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε μια πολύ καλή απόφαση που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά και ίσως βρεθούν και νέες λύσεις για να ξεπεράσουμε τις κληρονομίες του παρελθόντος. Θα ήθελα να, απα... να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κ. Μουρ. Ίσως σε κάποιες χώρες, όπως και στη Γερμανία, να μην συνειδητοποιούν οι πολίτες ε, ε, ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις ε, προμήθειες. Όμως σε άλλες χώρες, όπως και στη δικιά μου, συνειδητοποιούν οι πολίτες ότι η οικονομική κρίση την οποία ε, ζούμε τώρα οφείλεται στις ε, ε, στα προβλήματα και στις, ε, ε, τα οποία δημιούργησαν οι αγορές ας πούμε υποβρυχίων από την, από την Γερμανία και στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα λοιπόν οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει συμβάσεις, διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς σεβόμαστε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και ούτως ή άλλως αυτού του είδους τα συμβόλαια και συμβάσεις διαφθοράς αυτού του είδους ε, τις διατάξεις ε, ε, παραβιάζουν γιατί εδώ στα offsets στις δημιουργούνται τα προβλήματα και μιλάμε και για ιδιωτικές επιχειρήσεις εδώ, για ναυπηγεία και Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το κράτος, διότι το κράτος ε, συνάπτει αυτές ε, τις συμβάσεις. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η διαφθορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ε, είναι η διαφθορά των κρατικών υπαλλήλων και το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο έθιξε πρώτο το πρόβλημα αυτό, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία για τις κρατικές προμήθειες. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί στο κάτω-κάτω και τα χρήματα χρειαζόμαστε και θα πρέπει και οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο. Δεν τα δαπανούμε έτσι, ε, τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργηθούν οι ικανότητες οι οποίες έχουμε ανάγκη. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ ε, για τι εισηγήσει του και το έργο τους. Αυτές οι πληροφορίε πιστεύω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμε για τη δική μα έκθεση ιδία πρωτοβουλία ε, για το τις επιπτώσεις ε, των δημοσιονομικών περικοπών στα κονδύλια στην άμυνα των κρατών μελών. Και τις πληροφορίες που μας δώσατε ήταν πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωσή μας, λίγη ακρόασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.